Να ξεκινήσουμε, αγαπητοί συνάδελφοι. Είναι 3 ε, και τέταρτο. για τις ανακοινώσεις του Πρόεδρου, επειδή είχαμε κάποια προβλήτα γεγονότα, ε, δεν μπορεί να είναι Πρόεδρος ο κ. Μπρόκ. Ε, έτσι λοιπόν, σας ζητά να διαβάσω τη συγγνώμη του. Μας, μου ζητά να διαβάσω τη συγγνώμη του σε σχέση με το σημείο 5 για την ΚΕΠΑ. Ε, αυτό το σημείο θα το αναβάλουμε την ετήσια έκθεση λοιπόν για την ΚΕΠΑ. Θα περάσουμε λοιπόν στο ετήσιο πρωτόκολλο για ε, την συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Ισραήλ σχετικά με την αξιολόγηση της συμμόρφωσης και την αποδοχή βιομηχανικών προϊόντων. Η εισηγητρά για τη δική μας γνωμοδότηση από την ΑΦΕΤ είναι η συνάδελφος Δεκέισερ, που είναι εδώ παρούσα. Και έχουμε κατόπιν ε, μία γνωμοδότηση ΙΛΤΑ που έχει αναλάβει ο συνάδελφος Β. Μορένη. Σας υπενθυμίζω προθεσμία για τις τροπολογίες είναι 29 Μαρτίου στις 12 το μεσημέρι. Και σα θυμίζω ότι η ΑΦΕΤ ήδη έχει συζητήσει το εν ζήτημα βάσει ενός εγγράφου εργασία που παρουσιάστηκε από την εισηγήτρια τον προηγούμενο μήνα. Το έγγραφο το οποίο έθετε μια σειρά ερωτηματικών σε σχέση με την καταλληλότητα, τη σκοπιμότητα κύρωσης της συμφωνίας. Ε, ο εισηγητής στην ΙΝΤΑ μάλλον περιουσίασε μία πρόταση για μία ενδιάμεση έκθεση που ζητά το υνοπάγωμα της συμφωνίας για μία περίοδο δύο ετών. Και να σας θυμίσω ότι στην Επιτροπή συζητήσαμε την πρόταση της εισηγήτριας να ζητηθεί μία γνωμοδότηση της νομικής υπηρεσίας και ότι το διευρυμένο Προεδρείο ενέκρινε το αίτημα αυτό. Αυτή τη γνωμοδότηση την έχετε στη διάθεσή σας στο παράρτημα. Έτσι λοιπόν, στο σημείο αυτό θα δώσω το λόγο στην εισηγήτρια. Παρακαλώ κύριε Ντεκέισερ. Ε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε Αναφέρατε την ε, έκθεση στην Επιτροπή Ίντα, την οποία ε, συνέταξε ο συνάδελφος Βιτάλ Μορέιρα. Είναι ενδιαφέρον να διαπιστώσουμε ότι η έκθεση αυτή είναι αιτιολογημένη ε, από πολιτικές σκοπιμότητες ενώ μιλάμε για μια επιτροπή διεθνούς εμπορίου. Πρέπει λοιπόν εμείς που είμαστε η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων να συζητήσουμε και για την ουσία, για την πολιτική. Δεν μπορούμε δηλαδή να αφήσουμε την πολιτική ε, σκοπιά στην ε, διάθεση της Επιτροπής Ίντα. Και γι' αυτό πολύ σύντομα θέλω να αναφερθώ στο πολιτικό πλαίσιο αυτής της ε, συμφωνίας. Μετά θα σας πω τα αποτελέσματα της νομικής γνωμοδότησης, της θέσεις μου σαν εισηγητή και στο τέλος την τοποθέτηση της πολιτικής μου ομάδος σχετικά με το πολιτικό θέμα και ε, τα ανθρώπινα δικαιώματα που πρέπει ε, να χαρακτηρίζουν την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και την συνεκτική αντιμετώπιση της, το θέμα αυτό μας δημιουργεί προβλήματα, διότι για οποιοδήποτε προβλήματα και να συζητήσω, δηλαδή είτε μιλάμε για τις απικίες στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, είτε για ε, την κατάσταση στην, ε, ε, ε, στην πέρα όχθη του Ιορδάνη, το θέμα της Γάζας και τόσα άλλα βλέπουμε ότι υπάρχουν ε, τεκμηριωμένα θέματα τα οποία είναι αρκετά οξέα κατά τρόπον ώστε να έχουμε εκθέσεις των εκπροσώπων μας ε, από πέρυσι το χειμώνα για τις απικίες στη Δυτική Όχθη και στην ε, όχθη πέραν του Ιορδάνη και ε, τα σχόλια αυτά δεν προέρχονται από εμένα αλλά από ερευνητές οι οποίοι σήμερα καλούνται να διευκρινίσουν τα θέματα αυτά αλλά τα γεγονότα είναι δυστυχώς ε, απαράλλακτα διότι ε, στο, στην περιοχή Γάμα αυτή την οποία ονομάζουμε περιοχή Γάμα υπήρχε στην, προηγούμενη καταμέτρηση αριθμός 1.200 απίκων ενώ τώρα υπάρχουν πέραν των 3.000 Παλαιστινίων στη ζώνη αυτή. Στη δυτική ε, όχθη υπάρχουν 3.000 Ισραηλινοί άπικοι και ενώ υπάρχουν 120 ε, ε, επίσημες απικίες υπάρχουν και 100 ανεπίσημες διαθέσιμες, άρα σύνολο 3.000. Και με αυτόν τον τρόπο δεν είναι δυνατόν να ε, μπορέσουν να συμβιώσουν δύο κράτη ε, βάσει της γραμμής διαχωρισμού του 1967 και εκεί βασίζεται ε, η διεθνής και ευρωπαϊκή πολιτική μας η οποία κινδυνεύει για το θέμα της ειρήνης βάσει δύο κρατών βάσει μίας συνοριακής γραμμής η οποία σήμερα αμφισβητείται ε, και από τις δύο απικίες. Υπάρχουν όμως και άλλα προβλήματα. Και όλο αυτό το πολιτικό πλαίσιο οδηγεί στο ότι τώρα να συμφωνήσουμε με το πρωτόκολλο αυτό είναι σαν να δώσουμε ένα ενοχλητικό πολιτικό σήμα ότι το Ισραήλ στο θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ε, συνεκτικότητας της πολιτικής μας επ' αυτού μπορεί να αποτελέσει εξαίρεση το οποίο να απευχόμαστε. Και ε, γι' αυτό δεν μπορούμε αυτό το θέμα να το θίξουμε στην Επιτροπή ε, Εξωτερικών Υποθέσεων μέσω μίας γνωμονοδοτήσεως. Μπορούμε να δεχθούμε, να απορρίψουμε, αλλά να δώσουμε ένα μήνυμα. Και όλοι οι συνάδελφοι πρέπει να αντιληφθούν ότι το μήνυμα απευθύνεται στο Ισραήλ αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο, σε όλη την Ιφίλιο και ιδιαιτέρως στις χώρες της Αραβικής Ανοίξεως, τις οποίες ζητούμε αυτή τη στιγμή έντονα να σεβαστούν τα ανθρώπινα δικαιώματα στην μετάβαση προς τη δημοκρατία. Υπάρχει δηλαδή ένα σοβαρό πρόβλημα το οποίο δεν μπορούμε να αγνοήσουμε. Προτού ασχοληθώ με την νομική πτυχή έχω άλλη μία παρατήρηση διότι μου είπαν κυρία Κάιζερ εδώ μιλάμε για φάρμακα και συγκεκριμένα για φάρμακα τα οποία ενδιαφέρουν πάρα πολύ όλες τις χώρες μας, διότι το Ισραήλ είναι πρωτοπόρος στο χώρο της φαρμακευτικής και μέσα στους δέκα πρώτους εις ε, το διεθνές ε, πλαίσιο και στον, ε, το, στην κορυφή στον τομέα των γενοσύμων που ενδιαφέρουν την ευρωπαϊκή κοινωνική ασφάλιση. Άρα εγώ από τη μια μεριά μεν ας υπογράψω και να τα αποδεχτώ αλλά δεν καταλαβαίνω τότε γιατί στον μπλόκο της Γάζας ε, τα φάρμακα απετέλεσαν ένα όπλο πολέμου και ο προσωρινός ε, μηχανισμός που καταρτήσαμε για την Γάζα αναφερόταν καταρχήν, από τα, ε, καταρχήν στα φάρμακα υιοθετήθηκε από την Παγκόσμια Τράπεζα που χρειάστηκε ένα χρόνο για να διοχετεύσει φάρμακα στη Γάζα. Γιατί μου λέγουν τώρα ότι δεν υπάρχουν επαρκή φάρμακα στη Γάζα. Γιατί δεν μπορούμε να θεραπεύσουμε το 30% της αυξήσεως περιπτώσεων λευχαιμίας οι οποίες οφείλονται στους βομβαρδισμούς με ε, αποπλουτισμένο ουράνιο κατά τους βομβαρδισμούς. Θα ήθελα λοιπόν να δω την οργάνωση ΤΕΒΑ να εισέλθει πιο γρήγορα στην εσωτερική αγορά αν ήξερα ότι θα μπορούσε συγχρόνως να προσχωρήσει και πιο εύκολα στην Παλαιστινιακή αγορά και στη Γάζα. Δεν θέλω να μου λέγουν ότι η ιατρική δυστυχώς δεν χρησιμοποιείται ή στη διαμάχη μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστίνης διότι βεβαίως χρησιμοποιείται και πρέπει να μιλήσουμε καθαρά και ανοιχτά. Οι ομάδες μας ε, είναι διαχωρισμένες ε, η δικιά μου λιγότερο από άλλες διότι ορισμένοι θεωρούν ότι το Ισραήλ λόγω του παρελθόντος λόγω της ιστορίας η οποία ήταν τρομερή για τους Εβραίους στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο αξίζει περισσότερη προστασία και λόγω της ασφαλείας του η οποία κινδυνεύει. Και ορισμένοι μας λέγουν δεν μπορούμε να σας ακολουθήσουμε γιατί θα ερμηνευθεί σαν μια κίνηση κατά του Ισραήλ. Εγώ προσωπικά δεν δέχομαι αυτό το επιχείρημα αλλά σημειώνω ότι στην πολιτική μου ομάδα ορισμένοι ακολουθούν αυτό το σκεπτικό γιατί έχουν ένα εθνικό πλαίσιο που διαφέρει από το Βέλγιο και υπάρχουν παρεφερές καταστάσεις σε διάφορα κράτη. Γι' αυτό και ήθελα σε αυτή τη γνωμοδότηση ο καθένας να μπορέσει να βρει μία θέση που να τον αντιπροσωπεύει. Η θέση μου δηλαδή δεν είναι ούτε ναι ούτε όχι. Αυτό θα γίνει μέσω των τροπολογιών και είμαι σίγουρη ότι θα έχουμε και θετικές και αρνητικές πολιτικές τροπολογίες ακόμη και στην πολιτική μου ομάδα. Μπορώ να σας το ανακοινώσω. Αλλά σαν συμβιβαστική λύση θα βασιστώ στο νομικό θέμα. Και το νομικό θέμα όπως γνωρίζετε είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και η διεθνής κοινότητα αρνείται να εισέλθει στην ευρωπαϊκή αγορά αριθμός προϊόντων των απικιών τις οποίες δεν αναγνωρίζουμε ε, σαν ε, ε, Ισραηλινή επικράτεια και Ισραηλινά εδάφη. Ορισμένοι μου λέγουν ότι βεβαίως θα μπορούσαμε ενδεχομένω απλώς να πούμε ότι αν από τη μία πλευρά το Ισραήλ αναγνωρίσει τις απικίες ότι είναι μέρος της επικράτειάς του, οι Ευρωπαίοι όπως κάναμε και στο παρελθόν με το Ισραήλ ε, μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι δεν θέλουμε τις απικίες αυτές και ε, ε, ε, έχουμε διάφορες περιπτώσεις όπως η περίπτωση Μπρίτα η οποία δεν μας επιτρέπει να εισάγουμε προϊόντα των απικιών. Οπότε εμείς θα πρέπει να βρούμε ένα τρόπο να το αποφύγουμε και να το κλείσουμε εάν θέλουμε να προωθήσουμε αυτό το πρωτόκολλο. Εάν λοιπόν υπάρχει διατύπωση του παρελθόντος πρέπει να αναγνωρίζουμε ότι πρόκειται για ένα σουρωτήρι. Δεν μπορεί κανείς να ζητήσει από τελωνιακούς να πάνε, που είναι ανύπαρκτοι να πάνε να ελέγξουν την κατάσταση. Στη συμφωνία λοιπόν αυτή το Ισραήλ θα είναι αυτό το οποίο θα πιστοποιεί τα φάρμακα της δικής του επιλογής που θα συμμορφώνονται στα ευρωπαϊκά κριτήρια και στην ΆΤΑ το Ισραήλ θα κυριαρχήσει της κατάστασης και για τα προϊόντα και τα Ισραηλινά και των Παλαιστινίων και του Λιβάνου και των Επίκων και ε, της Δυτικής Όχθης του Ιορδάνη θα ελέγχει την κατάσταση ελέγχοντας στην ε, είσοδο μεγάλου αριθμού φαρμάκων στην ευρωπαϊκή αγορά και αν εισέρχονται στην ε, ε, στην αγορά του Ισραήλ θα εισέρχονται και στην Ευρώπη. Πράγμα που περιπλέκει ακόμη περισσότερο την κατάσταση αυτή των επίκων. Γι' αυτό και δεν θα παρουσιάσω την κατάσταση αυτή τώρα. Συμβουλεύτηκα νομικούς, τη νομική υπηρεσία, καθηγητές στο Πανεπιστήμιο των Βρυξελών και προτείνω εάν, και λέγω εάν, συνενέσουμε σε αυτό το πρωτόκολλο είναι ε, τουλάχιστον ε, το δικό μου συμπέρασμα αλλά θα υπάρξουν τροπολογίες. Εάν κάποτε δεχθούμε αυτό το πρωτόκολλο θα χρειαστεί ε, μία εξέταση και έκθεση η οποία θα προβλέψει ορισμένες προσθήκες και διευκρινήσεις όπου θα λέγεται ότι προϊόντα τα οποία προέρχονται από εδάφη των οποίων η κυριαρχία αμφισβητούνται δεν θα αποτελέσει αντικείμενο αυτού του παρατήματος. Πράγμα το οποίο επιτρέπει να πούμε ότι το παράρτημα του πρωτοκόλλου δεν θα καλύψει μόνο τα προϊόντα των επίκων αλλά και της Βορείας Κύπρου, της τουρκοκρατούμενης περιοχής, της Αυκασίας και άλλων δηλαδή δεν θα μπορεί κανείς να δεχθεί στην Ευρώπη και να εισάγει στην Ευρώπη φάρμακα που έρχονται από το Ισραήλ και ε, προέρχονται από αμφισβητούμενα εδάφη. Είναι μία δυνατότητα η οποία μπορεί να παρουσιαστεί στην ενδιάμεση αυτή έκθεση της Επιτροπής Ίνταμ και ε, πιστεύω ότι εφόσον θα υπάρξει μία προκαταρτική συμφωνία με ορισμένες επισφυλάξεις θα ικανοποιηθούν οι περισσότεροι. Σας παρακαλώ να καταλήξετε. Καταλήγω κύριε Πρόεδρε, δεν πρέπει να αφήσουμε την ίντα να διατυπώνει πολιτική αντιμών. Εμείς πρέπει να διατυπώνουμε την ε, πολιτική σε αυτό το σημείο για πέντε λεπτά. Το λόγο έχει ο κύριος Ιγνάσιο Πάρα από τη νομική υπηρεσία του Κοινοβουλίου. Μικρόφωνο παρακαλούμε. Θα είμαι σύντομος. Μοιράστηκε η γραπτή γνωμοδότηση, δεν θα επαναλάβω τόσο έλεγονται εκεί, απλώς ε, θα σας πω ποιο είναι το πλαίσιο, δηλαδή σε ποιο θα σκεπτικό μας τέθηκε και θα επικεντρωθούμε στην ερμηνεία του άρθρου 9. Σε ό,τι αφορά το πλαίσιο, αυτό το πρωτόκολλο θα, θα προσαρμοστεί στην Συμφωνία Σύνδεσης με το Ισραήλ το 2000. Αυτή η συμφωνία είναι ένα πρωτόκολλο τεχνικού χαρακτήρα ο στόχος του πρωτοκόλλου αυτού είναι να εξελίψει τα τεχνικά εμπόδια για την εμπορία των βιομηχανικών προϊόντων. Και ένα από τα μέσα του για την εξάλληψη των εμποδίων είναι ο διορισμός, ο καθορισμός αρμόδιων αρχών και από τις δύο πλευρές και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο Ισραήλ που να ελέγχουν τη συμμόρφωση με το ισχύον δίκαιο των προϊόντων που ε, μπορεί να μπουν στην αγορά. Πρόκειται για μια διαδικασία που υπάρχει και είναι παρόμοια με αυτή που υπάρχει στο ιστορικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης μεταξύ των κρατών μελών δηλαδή. Σε ό,τι αφορά το άρθρο 9, το άρθρο αυτό προβλέπει στη συγκεκριμένη περίπτωση ότι το Ισραήλ ε, αποστέλει στο άλλο μέρος, δηλαδή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τον καθορισμό μιας αρμόδιας αρχή για μια συγκεκριμένη επικράτεια. Το άλλο μέρος, ε, δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση, στο δικό μας παράδειγμα, οφείλει να επιβεβαιώσει γραπτός ε, αυτό το διορισμό. Και αυτό λέγεται στο άρθρο 9. Έτσι λοιπόν, καταρχήν έχουμε γραπτό καθορισμό μια αρμόδια αρχή για μια συγκεκριμένη επικράτεια και στη συνέχεια από την πλευρά τη Ευρωπαϊκή Ένωση θα γίνει γραπτή επιβεβαίωση αυτή του διορισμού. Ό,τι αφορά τώρα την επιβεβαίωση ή όχι από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, αυτό είναι ευθύνη της Κομισιόν κατά την ε, εκτέλεση του πρωτοκόλου. Το θέμα λοιπόν ε, των εδαφών που είναι υπό Παλαιστινική δίκηση από το 1967, αν τυθόταν θα ήταν στο πλαίσιο αυτό. Έτσι λοιπόν η Κομισιόν είναι αυτή που θα διαχειριστεί μια τέτοια κατάσταση. Αυτή θα είναι αρμόδια. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το σημείο έχουμε το κατάλογο των συναδέλφων που έχουν ζητήσει το λόγο. Να ξεκινήσουμε από τους κοιόδης εισηγητές και κατόπιν ε, της παρέμβασης των συναδέλφων από το Ευρωπαϊκό θα δώσουμε το λόγο και στον εκπρόσωπο της Κομισιόν για να απαντήσει. Η κυρία Γιαννάκου καταρχήν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, άκουσα με προσοχή την εισηγήτρια, την κυρία Ντεκάιζερ και επίσης μελέτησα την νομική γνωμοδότηση η οποία δόθηκε και της οποίας περίληψη μας ανέφερε ο ε, εκ μέρους της νομικής υπηρεσίας εδώ παρών. Ε, καταρχήν ε, να σημειώσω ότι από πλευράς νομικής δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα διότι η γνωμοδότηση είναι πάρα πολύ σαφής. Η άποψη του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος κύριε Πρόεδρε είναι αντίθετη από την άποψη της εισηγήτριας. Θεωρούμε ότι η συμφωνία αυτή πρέπει να γίνει όχι μόνο γιατί είναι προς όφελος και των δύο πλευρών αλλά και της Ευρώπης διότι πράγματι το Ισραήλ είναι από τις χώρες ε, που στον ερευνητικό τομέα και στην παραγωγή φαρμάκων βρίσκονται σε πάρα πολύ ψηλό επίπεδο ε, όχι μόνο διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει σχέσεις με πάρα πολλές τρίτες χώρες που φυσικά έχουν παρόμοια προβλήματα αλλά στην προκειμένη περίπτωση δεν ζητούμε να αγνοηθεί ε, το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει αναγνωρίσει τα εδάφη τα οποία έχουν καταληφθεί από το 1967 διότι η νομική γνωμοδότηση της ε, ε, νομικής υπηρεσίας μας παρέχει την ευχέρεια είτε ορίζοντας από την πλευρά του Ισραήλ τις αρχές οι οποίες είναι υπεύθυνες και έχουν την αρμοδιότητα με τον ορισμό ταυτόχρονα της περιοχής την οποία καλύπτουν είτε με τη δεύτερη λύση την οποία προτείνει η νομική γνωμοδότηση αυτή ε, αποκλείοντας τις συγκεκριμένες περιοχές. Έχω την εντύπωση ότι το να ζητήσουμε από την αρμόδια επιτροπή που είναι η ΙΝΤΑ να καθυστερήσει αυτήν την υπόθεση ή να κάνουμε ένα interim report ε, φοβάμαι κύριε Πρόεδρε ότι δεν θα ωφελήσει ούτε την Ισραηλινο-Παλαιστινιακή ε, σύγκρουση και διαμάχη. Αν επρόκειτο να προσφέρει αυτό κάτι επί της ουσίας ε, στο να λήξει το πρόβλημα αυτό το οποίο κρατάει πάρα πολλές δεκαετίες τότε θα σας έλεγα ναι, να ακολουθήσουμε την εισηγήτρια. Εισηγούμε λοιπόν να ζητήσουμε από την Επιτροπή Ίντα ευθέως ε, να συντάξει έκθεση θετική για, ε, για τη συμφωνία αυτή ε, σχετικά με τα βιομηχανικά προϊόντα, στην προκειμένη περίπτωση τα φάρμακα, ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ισραήλ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Ο κύριος Νταφ. Uh, Πρόεδρε, Φυσικά και συμφωνώ με την κυρία Ντεκάιζερ για το ότι το θέμα αυτό είναι ιδιαίτερα πολιτικό. Η νομική υπηρεσία μας το παρουσίασε σαν ένα τεχνικό ζήτημα. Εγώ δεν συμφωνώ. Δεν συμφωνώ ότι είναι τεχνικό. Δεν είμαστε αφελείς, δεν είμαστε αφελείς και γνωρίζουμε ότι όλα όσα έχουν να κάνουν με την φύση των σχέσεών μας με το Ισραήλ είναι κυρίως πολιτικά θέματα. Έχουν πολιτική διάσταση. Και γι' αυτό ως Κοινοβούλιο καλούμεθα να αποφασίσουμε. Συμφωνώ με την κυρία Γιαννάκου για το ότι δεν έχουμε να κερδίσουμε τίποτα μην παίρνοντας μια δύσκολη πολιτική απόφαση. Ως Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων πρέπει να αναρωτηθούμε κατά πόσο συμφωνούμε ή διαφωνούμε με την συμφωνία. με το τι επιπτώσεις θα έχει στις σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το Ισραήλ. Εγώ θα ήθελα να μπορούσα να συζητήσω αυτό το θέμα με την ύπατο εκπρόσωπο. να, ενημερωθεί, να ενημερωθούμε μάλλον από τους διπλωμάτες μας επίσης, κάτι το οποίο πιστεύω ότι είναι ζωτικής σημασίας. Υπάρχει βέβαια ένα νομικό ζήτημα, διότι το Ισραήλ, κατά τη γνώμη μου, δεν μπορεί να δεσμευτεί να μην εφαρμόσει κατά από τους όρους της συμφωνίας την συμφωνία αυτή στα κατεχόμενα. Συνεπώς, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα βρεθεί σε μια πολύ ατυχή κατάσταση. Νομικά μιλώντας και σε μια παράνομη βασικά κατάσταση. Για να συνοψίσω λοιπόν, η ομάδα των φιλελεύθερων είναι υπέρ μιας απόφασης, να μην καθυστερήσουμε δηλαδή, να μην καταλήξουμε σε μια έτσι αμφίσιμη πρώτη έκθεση. Όσον αφορά την ουσία τώρα της πολιτικής απόφασης, τελικά θα πρέπει να περιμένουμε και να δούμε τι απόφαση τελικά, προς ποια κατεύθυνση τελικά θα θελήσει να πάει η ομάδα. Πάντως για μένα, ειλικρινά, θα ήταν να αντιταθούμε στην συμφωνία. Λοιπόν, τρίτο σκιώδη, τρίτη σκιώδη μάλλον, η κυρία Νίλσεν. Παρακαλώ. Je pense... Πιστεύω πως και η κυρία Ντεκίζερ. Όχι μόνο δεν βλέπουμε ε, κάνει ένα θετικό βήμα από το Ισραήλ να πληρώσει τις υποχρεώσεις που το έχουν υπευληθεί δυνάμει του διεθνούς δικαίου, αλλά αντίθετα βλέπουμε κάποια σημάδια κλιμάκωσης, ε, δημιουργία νέων επικισμών, ε, προσάρτηση γεών και του ύδατος, ζωτικών δηλαδή πόρων και επίσης υπενθυμίζω το θέμα ε, του νερού και της ε, χρησιμοποίησης ε, του νερού υπέρ των επίκων και εις βάρος των Παλαιστινίων. Στις 19 Μαρτίου είχαμε μάλιστα και μία έκθεση του ΟΗΕ που έκρουσε τον κόδωνα του κινδύνου για το θέμα αυτό. Ε, κυρία Ντεκέιζερ μίλησε για την αρπαγή των γιών και ξέρετε ότι ο ΟΗΕ θέλει να κάνει μία επίσημη έρευνα για τον αντίκτυπο ε, της συνεχής κατασκευής κατασκευής, της συνεχούς κατασκευής των νέων επικισμών ε, στη Δυτική Όχθη και ξέρετε ότι ο αριθμός των επίκων έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία έτη. Επίσης ε, θα ήθελα να αναφερθώ στην ενέκθεση των ε, επικεφαλής των αποστολών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, που στην έκθεση αυτή μεταξύ άλλων μας συμβουλεύουν να κάνουμε μια πραγματική ενημερωτική εκστρατεία στην Ευρώπη κυρίως στις επιχειρήσεις, να απευθυνθούμε στις επιχειρήσεις και να τις παρατηρούμε να μην επενδύουν στους ενεργοεπικισμούς. Πιστεύω λοιπόν ότι αυτό το σημείο είναι σημαντικό να το θυμόμαστε και από ε, την επιχείρηση ε, του Ισραήλ ε, στη Λωρίδα της Γάζας. Έχουμε πολλά σχέδια που χρηματοδοτήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε ένα κατάλογο εδώ που χρηματοδοτήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα οποία καταστράφηκαν από το Ιόνιο στρατό, πρόκειται για ταξαμενέ νερού, πρόκειται για καταβλισμού, πρόκειται για καταφύγια ή για μια φωτοβολταϊκή εγκατάσταση ε, Πρόκειται για ε, πολύ σημαντικέ επενδύσει τη Ευρωπαϊκή Ένωση ε, στην ζώνη αυτή που καταστρέφονται από τον Ισραηλινό στρατό. Πιστεύω λοιπόν από πολιτική σκοπιά πραγματικά αυτό μα κάνει να αναρωτιόμαστε και για μένα είναι προφανή τα πράγματα. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε με τον τρόπο αυτό και να προποιούμαστε ότι τα πράγματα συμβαίνουν ε, κανονικά ομαλά με το Ισραήλ και σίγουρα δεν υπάρχει καμία εγγύηση τη συνεργασιμότητα στην Ευρώπη ξέρουμε ότι έχουμε πάρα πολλές ενώσεις στη Γαλλία, στην Ευρώπη. Μας απέδειξαν ότι ε, υπήρχε εισαγωγή προϊόντων από τους επικισμούς και δεν έφεραν ε, τις ε, κατάλληλες επισημάνσεις. Και νομίζω λοιπόν ότι δεν υπάρχει σεβασμός της συμφωνίας μεταξύ Ισραήλ και Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν υπάρχει καμία εγγύηση σε ό,τι αφορά την εφαρμογή του πρωτόκολλου Τώρα, για το νομικό τμήμα, άκουσα τι υπόθηκε ό,τι αφορά την γνωμοδότηση της νομικής υπηρεσίας. Το πρόβλημα είναι ότι η Κομισιόν είναι αυτή η οποία θα πρέπει να διασφαλίσει ότι ε, υπάρχει σεβασμός του δικαίου. Εμείς δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό στο Κοινοβούλιο. Εμείς έχουμε κάποιες πολιτικές απόψεις σε ό,τι αφορά την πολιτική του Ισραήλ και την κατοχή των Παλαιστινιακών εδαφών. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι σαφή τα πράγματα. Εδώ ως μέλη του Ευρωπαϊκού Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, είμαστε σε μια επιτροπή και ο ρόλο μα είναι για να λάβουμε μια πολιτική απόφαση και όχι τεχνικού χαρακτήρα απόφαση, όπω μα κάνουν κάποιοι να σκεφτούμε. Και επίση από τους ε, γιατρού, του Γάλλου που εργάστηκαν στη Γάζα, ξέρω ότι δεν υπάρχουν αρκετά φάρμακα και ιατρικό υλικό στη Γάζα για την ε, θεραπεία των τραυματιών, γιατί είχαμε 1.400 ε, νεκρούς από την επιχείρηση του Βίλαν. έχουμε και πάρα πολλά άτομα που έμειναν ανάπηρα και δεν υπάρχουν αρκετά φάρμακα για αυτού. Έτσι λοιπόν θεωρώ ότι είναι σοκαριστικό να σκεφτόμαστε ότι μπορούμε να υπογράψουμε αυτή τη συμφωνία που αφορά απλώς φάρμακα ε, όταν γνωρίζουμε σε ποια υγειονομική κατάσταση βρίσκεται ο πληθυσμό στην Παλαιστίνη τόσο στη Γάζα όσο και αλλού. Και θέλω να επιμείνω και στι γυναίκε, οι οποίε βρίσκονται σε ε, άθλιες συνθήκε σε ό,τι αφορά τη μητρότητα. Ο συνάδελφος Σίβιτς παρακαλώ έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Είναι δεύτερη φορά που συζητάμε ένα θέμα το οποίο φαίνεται ε, καταρχήν εύκολο αλλά είναι πολύ φορτισμένο συγκινησιακά διότι ε, πρέπει να μην έχουμε πλέον αμφιβολίες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ε, ελαφρά καρδιά να μπορέσουμε και να σεβαστούμε την νομοθεσία στην οποία βασίζεται η Συμφωνία Συνδέσεως, να μην υπάρχει δηλαδή παραβίαση της νομοθεσίας εάν εγκρίνουμε αυτό το πρωτόκολλο και να μην επιτρέψουμε να παραβιαστεί αυτή η νομοθεσία κάπου αλλού μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και του Ισραήλ. Η κυρία Ντεκάιζερ μας είπε ότι είναι ένας πολιτικός χώρος εδώ και τα θέματα πρέπει να συζητούνται όταν αποφοραούν το εμπόριο στην Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Θέλουμε να αναρωτηθούμε εάν θέλουμε να τιμωρήσουμε το Ισραήλ και αν ναι πρέπει να δούμε για ποιο λόγο, για την έλλειψη ειρήνης στη Μέση Ανατολή, διότι αν θέλουμε γι' αυτό να τιμωρήσουμε το Ισραήλ δεν είναι ο μόνος υπέτειος, υπάρχουν και άλλοι υπέτειοι στη Μέση Ανατολή για την ισχύουσα κατάσταση. Θέλουμε να τους πιέσουμε διότι υπέγραψαν μία τέτοια συμφωνία συνδέσεως. Δεν νομίζω, διότι και άλλοι υπογράφουν τέτοιες συμφωνίες συνδέσεως. Ίσως λοιπόν είμαστε ε, καταπιεσμένη από την βία στην λωρίδα της Γάζας, από τους ανθρώπους ε, οι οποίοι υποφέρουν, αλλά δεν νομίζω ότι είναι ο τρόπος αυτός να εκτονωθούμε. Όταν λοιπόν παρακολουθώ τη συζήτηση αυτή, εκπλήσωμαι διότι υπάρχει μία διασύνδεση μεταξύ των φαρμάκων εις ε, την ε, ε, λωρίδα του Ισραήλ και των φαρμάκων που φτάνουν στην Ευρώπη. Δεν νομίζω ότι μιλάμε για τα ίδια φάρμακα. Δεν θα βοηθήσουμε τους κατοίκους της Γάζας τιμωρώντας το Ισραήλ με αυτόν τον τρόπο, διότι η αρχή αυτή είναι αυτή που διέπει την πολιτική μας γυτνιάσεως. Και υπάρχει κίνδυνος να αποδειχθούμε εδώ πολύ υποκριτές. Το Ισραήλ περιμένει δύο χρόνια, δεν νομίζω ότι χρειάζεται να περιμένει άλλα δύο. Συνάδελφοι, πρέπει να περιοριστείτε στις παρεμβάσεις σας τα δύο λεφτά, γιατί διαφορετικά δεν θα έχουμε αρκετό χρόνο για να ακούσουμε και τις απαντήσεις της ηχήτριας, ούτε της Κομισιόν. Δεν θα μας φτάσει ο χρόνος. Παρακαλώ, Μπράνερ, δύο λεπτά. Yes, thank you, Mr. President. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Αυτό που είναι σημαντικό είναι να έχουμε στο μυαλό μας ότι για δύο λόγους συζητάμε είτε την προσωρινή έκθεση είτε την αναβολή. Και νομίζω ότι και για την πρώτη περίπτωση πάλι έχουμε δύο λόγους. Πρέπει να καθορίσουμε κριτήρια πρώτα απ' όλα για το πότε θα πούμε εντάξει Οπότε λοιπόν θα συμφωνήσουμε. Και οι δύο λόγοι που ανέφερε η Βερονίκ και άλλοι είναι η σημερινή κατάσταση πραγμάτων στο Ισραήλ, εκεί που είναι η έπικη, πρόκειται για πολιτικό μήνυμα και άρα πρέπει να προσέξουμε ποια στοιχεία θα το δώσουμε. Και το άλλο είναι πώς θα διασφαλίσουμε ε, τι θα γίνει με τα προϊόντα αυτών. Συνεπώς πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί Και η ερώτησή μου προς τη Βερονίκη είναι εξή. Αν κάνουμε ενδιάμεση έκθεση, προσωρινή έκθεση, που η ομάδα μας το θέλει, τότε τι προτείνεται ως κριτήρια προκειμένου να φτάσουμε στο στάδιο που θα πρέπει να πούμε ναι ή όχι. Να μπορέσουμε να αποφασίσουμε δηλαδή. Ο κύριος Χουμπής, γιατί είναι σκιώδης εισηγητής. Τρία λεπτά έχετε ως σκιώδης εισηγητής. Okay. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θεωρώ ότι δεν μου δώσατε το λόγο με τη σειρά που θα έπρεπε ως τεχνικό θέμα και όχι πολιτικό. Ως τεχνικό θέμα. Εκ παραδρομής. Επειδή μπήκαμε σε αυτή την ορολογία. Θέλω να σας πω ότι ε, συμφωνώ με τις απόψεις που εξέφρασε η συγγήτριά μας. Το θέμα είναι πολιτικό. Αυτό είναι πολιτικό θέμα. Και νομίζω ότι εδώ πρέπει να, η Επιτροπή μας να αποφανθεί με βάση το δίκαιο και με βάση την ε, συμπεριφορά του Ισραήλ σε σχέση με το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων των Παλαιστινίων. Δυστυχώς, λόγω μιας γενικότερης ανοχής που εισπράττει το Ισραήλ, η κατάσταση επιδεινώνεται. Σημειώνω και εγώ για άλλη μια φορά ότι πριν λίγες μέρες, χτες μάλλον, το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι διακόπτει κάθε επαφή με το Συμβούλιο του ΟΗΕ σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα σε σχέση με απόφαση του Συμβουλίου του ΟΗΕ να ανοίξει διεθνή έρευνα για τους Ισραηλινούς επικισμούς και θα μπορούσε κανείς να αναφέρει και άλλα θέματα. Η ομάδα μας και εγώ προσωπικά η ομάδα μας έχει ενιαία θέση και πιστεύει ότι και είμαστε αρνητικοί για την ανάπτυξη του εμπορίου και για ενισχυμένες σχέσεις με το Ισραήλ ως αυτό συνεχίζει και παραβιάζει το διεθνές δίκαιο, τα δικαιώματα των Παλαιστινίων. Δεν θεωρούμε ότι το θέμα είναι τεχνικό, όπως αποφαίνεται η νομική επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα σας έλεγα εκ της εμπειρίας ανάλογων ή αντίστοιχων προβλημάτων στην περιοχή, πολλές φορές ή ορισμένες φορές πολιτικά ζητήματα ή θέσεις αρχών τείνουν να παρακάμπτονται με υποτίθεται τεχνικά προβλήματα και κυρίως με το θέμα του εμπορίου και των εμπορικών σχέσεων. Θέλω να πω ότι η λογική ότι δεν λύνουμε το πρόβλημα αλλά ενδεχομένως διευκολύνουμε στη συμμόρφωση του Ισραήλ ή οποιοδήποτε κράτος διευρύνοντας τις εμπορικές σχέσεις δεν έχει αποδειχθεί ότι είναι η κατάλληλη συνταγή. Και στην προκειμένη περίπτωση δεν νομίζω ότι πρέπει να πάμε προς, αυτό αυτή την κατεύθυνση. Επειδή αναφέρθηκε κάποιος ε, προηγούμενος ομιλητής, δεν νομίζω ότι με τη θέση αυτή ή όποιος εκφράζει μια τέτοια θέση, δηλαδή να αρνηθούμε την υπογραφή αυτού του πρόσθετου πρωτοκόλου, να προτείνει η δική μας Επιτροπή, ότι απλώς εκτονώνουμε την αλληλεγγύη μας προς τους Παλαιστινίους. Νομίζω ότι υπερασπιστόμαστε μια θέση αρχών, υπερασπιζόμαστε το ευρωπαϊκό δίκαιο και δεν πρέπει να δώσουμε κακό δείγμα χαλάρωσης ή ρήγματος μέσω μιας τεχνικής και άλλης υπόθεσης. Και τέλος, το επιχείρημα, επειδή ακούγεται και στη χώρα μου τελευταία, περί της πρωτοπορίας του Ισραήλ και στα φάρμακα, θυμίζει άλλες καταστάσεις και άλλες ας το πούμε προτεραιότητες δεν νομίζω πως πρέπει, πως πρέπει αυτές να μπουν στη δική μας γνωμοδότηση και να την χαρακτηρίσουν. Η πρότασή μας λοιπόν είναι να προτείνουμε να μην υπογραφεί αυτό το πρόσθετο πρωτόκολλο. Ευχαριστώ. Τέλειωσα κύριε Πρόεδρε. Τέλειωσα. Ευχαριστώ. Λοιπόν, πριν να συνεχίσουμε, ήθελα να υπογραμμίσω στον συνάδελφο ότι σας δώσαμε το λόγο τη στιγμή εντοπίσαμε την παρουσία σας γιατί δεν ήσασταν στον κατάλογο δεν θέλαμε να κάνουμε κάποια διάκριση απέναντί σας Παρακαλώ ο κύριος Έντριν, ευχαριστώ ναι, αυτό είναι όντω ε, πολιτικό ζήτημα. Υπάρχουν οι νομικέ πτυχές ε, και η νομική πτυχή είναι τεχνικό ζήτημα ίσως, αλλά είμαι σίγουρος ότι ό,τι και να αποφασίσουμε θα καλυφθεί με κατάλληλο τρόπο από νομική σκοπιά. Έτσι λοιπόν το καθήκον μας είναι να λάβουμε μια πολιτική απόφαση. Και το να μην λάβουμε καμία απόφαση δεν είναι κάτι σωστό. Θα έλεγα ότι η αναβολή δεν είναι πολιτική επιλογή και δεν είναι πολιτική επιλογή γιατί αυτή η αναβολή ποτέ δεν λύνει τα προβλήματα. Μάλιστα, ούτε μας βοήθησε να επιλύσουμε τα προβλήματα και αυτό το συγκεκριμένο πρόβλημα που έχω κατά νου, ούτε μας προσέφερε καλύτερη υποστήριξη για τη δική μας πολιτική στον υπόλοιπο κόσμο πρόσφατα ε, είχαμε μία διάσκεψη εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που μας έδωσε τη δυνατότητα να ακούσουμε ένα πυρογνώμονο που μας είπε ότι παρά το ότι η πολιτική μας στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, είναι ιδιαίτερα συνεπής, τα τελευταία χρόνια χάνουμε υποστήριξη εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι λοιπόν, ε, βεβαίως ε, πολλοί έχουν ε, διαφορετική άποψη για το πώς πρέπει να επιτευχθεί η ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή. Βεβαίως και έχουμε συμπόνια για τους ανθρώπους που υποφέρουν εκεί και έχω καταρχήν στο νόμο της Παλαιστινίους. Αλλά καθώς ε, δεν μπορούσαμε να αποκτήσουμε περισσότερη επιρροή στο παρελθόν, νομίζω ότι τώρα πρέπει να σκεφτούμε μια διαφορετική πολιτική, ιδίω αν θέλουμε να έχουμε περισσότερη επιρροή και να εμπλακούμε καλύτερα στο διάλογο με το Ισραήλ. Θα έλεγα, αν θα μπορούσε να είναι και το Ισραήλ. Χρησιμοποιεί, παραδείγματο χάρη, τα φάρμακα ω ε, όπλο ε, πολέμου. Ακριβώ γι' αυτό δεν πρέπει να το κάνουμε. Δηλαδή, να δώσουμε το μήνυμα ότι εμεί δεν είμαστε τέτοιοι άνθρωποι, δεν είμαστε τέτοιοι άνθρωποι, ούτε τέτοια ένωση που χρησιμοποιεί τα φάρμακα για αυτό το σκοπό. Και τελευταία πρόταση, Πρόεδρε, ότι σύμφωνα με τη συνθήκη τη Λισαβόνα, η Ένωση υποτίθεται ότι πρέπει να προωθεί τι δικέ τη αξίε. Ε, άρθρο 2, το συμφέρον της Ένωσης και την ασφάλεια των λαών, των πολιτών. Είναι πάρα πολύ δύσκολο πάντοτε στο δύο καλάθι να τα βάλουμε όλα και τα τρία αυτά. Νομίζω ότι προκειμένου να τα βάλουμε αυτά από κοινό αυτή τη στιγμή πρέπει να, κάνουμε, να λάβουμε μία απόφαση η οποία πρέπει να είναι και θετική. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η κυρία Αντρικίνε. Thank you, Mr. Chairman. Ευχαριστώ, συνάδελφοι. Πρέπει να ζητήσουμε από την Επιτροπή είτε να δώσει τη σύμφωνη γνώμη. Αυτά που συζητάμε σήμερα είναι θέματα που το Συμβούλιο και η Επιτροπή έχουν συζητήσει και συμφωνήσει πάνω σε αυτά εδώ και δύο χρόνια. Κάθε καθυστέρηση θα ζημιώσει την Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν θα βελτιώσει την επιρροή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή. Το Ισραήλ χρειάζεται ε, κάποια προνόμια. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία συνέταξε το κείμενο αυτό, λέει ότι άκα θα δημιουργήσει ωφέλη γιατί θα διευκολύνει την πρόσβασή μας σε αγορές. Επιπλέον, θα ενισχύσει τη συνεργασία μας στη Μέση Ανατολή. Εγώ θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι κάθε διευκόλυνση, είτε πρόκειται για την Ιορδανία, την Αίγυπτο, χρειάζεται συμφωνία από το Ισραήλ και έχει να υποφεληθεί από την προτιμησιακή μεταχείριση της συμφωνίας. Θέλω λοιπόν να υπογραμμίσω ότι η υπογραφή της δεν αναβαθμίζει τις εξωτερικές σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το Ισραήλ, Θέλω επίσης να προσθέσω ότι η συμφωνία αυτή είναι μέρος μιας περιφερειακής διαδικασίας που ξεκίνησε με τη διαδικασία της Βαρκελόνης για την εταιρική μεσογειακή σχέση. Είναι μια επιπλέον συμφωνία στην Συμφωνία Σύνδεσης Ευρωπαϊκής Ένωσης Ισραήλ και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής. Τώρα οι ανησυχίε μα όσον αφορά την εφαρμογή τη συμφωνία ε, στα κατεχόμενα εδάφη του παραβίαση των υποχρώσεων τη Ευρωπαϊκή Ένωση βάσει διεθνών ε, συμφωνιών και δικαίου, οι νομικέ υπηρεσίε απάντησαν σε αυτό. Ο ορισμός δεν μπορεί να είναι ε, διαφορετικός από ό,τι στην συμφωνία εταιρικής σχέσης. Έπειτα, ορισμός των εδαφών είναι θέμα εφαρμογής της συμφωνίας και δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι θέμα πάλι εφαρμογής και δεν απαιτεί τροποποίηση της συμφωνίας. Συνεπώς, πιστεύω ότι μπορούμε να προχωρήσουμε αντιμετωπίζοντας θετικά τη συμφωνία αυτή. Ευχαριστώ. Είχαμε την ευκαιρία να ακούσουμε στο διευρυμένο Προεδρείο τον Υπουργό Εξωτερικών της Παλαιστίνης μας εξήγησε το διέξοδο στο οποίο βρίσκεται η ειρηνευτική διαδικασία ως συνέπεια του πρωταγωνιστικού ρόλου της Αραβικής Άνοιξης και των εκλογικών διαδικασιών. Σε είπα και Ισραήλ εδώ, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο βρίσκεται απέναντι μια ευαίσθητη πολιτική απόφαση και προσπαθούμε να δούμε αν αυτό το πρόσθετο πρωτόκολλο στη Συμφωνία Σύνδεση πρέπει να ακυρωθεί ή όχι. Η προσωπική μου άποψη, Πρόεδρε, είναι ότι δεν πρέπει να μπλέκουμε το στόχο με την ουσία και δεν πρέπει να μπλέκουμε ε, τις σκιές ε, της εικόνας ε, με την ίδια την εικόνα. Θα πρέπει να κάνουμε μία, μία, ναι, μία πρόταση σε σχέση με το πολιτικό σκηνικό που κατά την άποψή μου θα έπρεπε να δώσει μία θετική γνώμη παρά τη στάση του Ισραήλ. Όμως νομίζω ότι πρέπει να λάβουμε υπόψη για κάτι που είπε η κυρία Ντεκάισερ και είναι σημαντικό ότι ούτε εμείς ε, θα πρέπει να επιτρέψουμε να εφαρμοστεί αυτή η συμφωνία στα εδάφη που κατέχει το Ισραήλ από το 67. Ίσως θα μπορούσαμε να βρούμε μία λύση συμβιβασμού που θα μπορούσε να διατηρήσει την αρχή που όλους μας συγκινεί και όπως ε, είπε και η κυρία Γιαννάκου θα μπορούσε να είναι σε αυτή τη γραμμή. Πιστεύω πάντως ότι πρέπει το θέμα αυτό να το δούμε ισορροπημένα και να λάβουμε υπόψη και την πολιτική διάσταση που κατέχει. Ευχαριστώ. Γκόμες. Γκόμες, παρακαλώ, κυρία Γκόμες, δύο λεπτά. Κύριε Πρόεδρε, αντιλαμβάνομαι τα επιχειρήματα τα οποία χρησιμοποιούνται και ιδίω την προσπάθεια που κάνει ο εισηγητής μας να βρει ε, μία συμβιβαστική λύση που θα συσπηρώσει το Κοινοβούλιο και θα επιτρέψει σε αυτή την πολιτική επιτροπή η οποία κάνει μία πολιτική αξιολόγηση να ακολουθήσει μία συνεκτική πολιτική με την ευρωπαϊκή νομολογία και Αλλά ε, και εγώ συμφωνώ με τη Βερονίκ Κάιζερ ότι ασχέτως των τεχνικών λεπτομεριών και είναι πολλές, το θέμα αυτό είναι ένα θέμα πολιτικής κρίσεως που αμφισβητείται και λαμβάνοντας υπόψη το τι γίνεται ε, και ε, τι κάνουν οι εταίροι μας δεν είναι μόνο οι Ισραηλινοί εταίροι μας δεν θέλουμε εδώ να τιμωρήσουμε το Ισραήλ αντιθέτως να ε, εμποδίσουμε το Ισραήλ να συνεχίσει να αυτοτιμωρείται τιμωρώντας τους Παλαιστινίους γιατί με τις πράξεις αυτές αυτές Ισραήλ αυτό τιμωρείται και γι' αυτό θα ε, υποβάλω μία τροπολογία αρνούμενη αυτό, δηλαδή πρέπει να γίνει μόνο μία πολιτική αξιολόγηση και να δούμε ε, τι, ε, πώς πρέπει να ερμηνεύεται η ευρωπαϊκή νομοθεσία όταν τα ανθρώπινα δικαιώματα έχουν κάποια σημασία. Κύριε Βάιντερ, ευχαριστώ. Καθώς ε, δεν έχω πολύ χρόνο για να σχολιάσω, δεν ε, θα ήθελα να επαναλάβω σε υπόθηκε προηγούμενες ομιλητέ. Ε, εγώ συμφωνώ απόλυτα με όσα υπόθηκαν από του κυρίου Σίβετ και Γιαννάκου. Περιέγραψαν πάρα πολύ καλά την κατάσταση και συμφωνώ και με τον κύριο Σαλαφράγκα και την κυρία Ντρικένε. Συμφωνώ με όλα όσα είπαν λοιπόν οι συνάδελφοι. Παρ' όλα αυτά θα ήθελα να επενθυμίσω κάποια πράγματα και να αναφέρω κάποιε ομοιότητε. Γιατί, αν παραδείγματο χάρη ακολουθήσουμε αυτή τη λογική και αν θέλουμε να επιλύσουμε όλα αυτά τα περιφερειακά προβλήματα με, το, με αυτό το πρόσθετο πρωτόκολλο, ε, τότε εκείνοι οι βουλευτέ που είναι κατά του πρωτοκόλλου αυτού θα έπρεπε να ψηφίσουν υπέρ του παγώματο όλων των εμπορικών συναλλαγών με την Αρμενία. Το ίδιο θα έπρεπε να γίνει δηλαδή και με την Αρμενία και με την Ρωσία πριν να λυθεί το πρόβλημα της Νότιας Οσετίας. Έτσι λοιπόν πρέπει να κάνουμε μια διάκριση μεταξύ των εμπορικών ε, σχέσεων που ευνοούν και τα δύο μέρη από τις πολιτικές σχέσεις. Και με το πρωτόκολλο αυτό δεν θα μπορέσουμε να λύσουμε όλα τα προβλήματα σε αυτή την περιοχή, τα οποία φυσικά και θα έπρεπε να λυθούν. Παρ' όλα αυτά, θέλω να απευθύνω μία έκκληση να εγκρίνουμε αυτή τη συμφωνία ΚΑ, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντική για όλη την περιοχή σας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Τάνοκ. Δύο λεπτά. Uh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η συζήτηση αυτή μου δίνει το συνέστημα του déjà vu. Είναι ξαναμασιμένο φαγητό. Έχουμε ξανακάνει αυτή τη συζήτηση. Οι θέσεις δεν έχουν μετακινηθεί καθόλου και έχουν σκληρύνει ε, μάλιστα αντιθέτως και ε, βλέπω ότι η Επιτροπή αυτή προσπαθεί να τιμωρήσει με κάθε τρόπο το Ισραήλ και στο θέμα της ΆΤΑ, του επιπρόσθετου πρωτοκόλου για τα φάρμακα, ακόμη και αν ε, μπορεί κανείς ε, να αγοράσει φθηνά και πολύ καλά φαρμακευτικά προϊόντα από το Ισραήλ. Άκουσα όλα τα πολιτικά σχόλια, τα, νομίζω ότι όλοι τα καταλαβαίνουμε, αλλά δεν βλέπω τώρα η καθυστέρηση να συνενέσουμε σε αυτό το πρωτόκολλο πρόκειται να βοηθήσει το λαό ή την κυβέρνηση του Ισραήλ και να πιστέψουν στην καλή πίστη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και την καλή διάθεσή του ε, προς το Ισραήλ. Γι' αυτό και νομίζω ότι τώρα πρέπει να αποφασίσουμε, όχι σε δύο χρόνια, και να συνενέσουμε κοινοβουλευτικά στο επιπρόσθετο πρωτόκολλο της ΆΤΑ και ε, έτσι πρόκειται να ψηφίσει και η πολιτική μου ομάδα επί του θέματος. Ευχαριστώ. Η συζήτηση τώρα μπήκε στην ουσία. Η πλειοψηφία των συναδέλφων ε, τοποθετήθηκαν, ε, είπαν την άποψή του ότι είναι πολιτικό και όχι τεχνικό το ζήτημα και εγώ δεν καταλαβαίνω σε ποια βάση μπορεί να υποβαθμιστεί και να παραγωνιστεί ως ένα ζήτημα ισονοσημασίας. Δεν μιλάμε μόνο για το Ισραήλ και την πολιτική του, μιλάμε για το διεθνές δίκαιο και για τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα. Αν εμείς λοιπόν σε αυτό το κοινοβούλιο υποφασίσουμε ότι στι εξωτερικέ εμπορικέ μα σχέσει δεν θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη τα ανθρώπινα δικαιώματα και άλλου παράγοντε. Δεν θέτουμε κανένα όρο. Αυτό είναι μία απόφαση. Αλλά αν αποφασίσουμε να θέσουμε κάποιου όρου και αν αποφασίσουμε ότι η ρησιμότητα είναι σημαντική και σε κάθε εμπορική συμφωνία με άλλε χώρε βάλουμε και αυτό το θέμα, θα πρέπει να είμαστε συνεπεί. Δεν μπορούμε να αλλάζουμε του όρου και τι προποθέσει ε, ανάλογα με τη χώρα ανάλογα με το μέγεθο τη χώρα ή την πολιτική σημασία τη χώρα Και το Ισραήλ είναι μια μικρή χώρα, αλλά είναι πολύ σημαντικό από πολιτική σκοπιά, για λόγους που όλοι του γνωρίζουν. Με τη συμφωνία αυτή λοιπόν δεν θα έπρεπε να κρύβουμε το πραγματικό πολιτικό πλαίσιο. Κατά την άποψή μου θα έπρεπε να απορρίψουμε τη συμφωνία. Γιατί ε, το Ισραήλ παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα και γιατί θα πρέπει να είμαστε συνεπείς ε, με το θέμα του μεγέθους των παραβιάσεων. Δεν είναι ε, αυτές οι παραβιάσεις όλες οι ίδιες, αλλά δεν μιλάμε για μια χώρα η οποία κατέχει εδάφη άλλης χώρας. Και μιλάμε για μια κατάφορη παραβίαση των ανθρωπινών δικαιωμάτων. Μιλάμε για πόλεμο πρέπει να είμαστε συνεπείς. Ε, πολλές φορές ε, καταδικάζουμε ε, μια μεγάλη χώρα για πολύ μικρές τις υπεραβίας ανθρωπίνων δικαιωμάτων και χρησιμοποιούμε διαφορετικά κριτήρια. Όμως δεν θα πρέπει να τα ξεχνάμε όλα αυτά όταν συζητούμε το θέμα του Ισραήλ και αυτής της συμφωνίας. Πολύ ωραία λέει ο πρόεδρος. Λάτφορτ, παρακαλώ. Συνάδελφος Λάτφορτ. Ευχαριστώ κυρία, κύριε Πρόεδρε συμφωνώ με ε, σχεδόν όλα τα σχόλια που παρουσιάστηκαν εναντίον της συστάσεως της κυρίας Δεκάιζερ και όπως είπε και ο κύριος εν ονόματι των φιλελευθέρων αυτό που χρειαζόμαστε είναι να καταλήξουμε σε μία απόφαση δηλαδή να προχωρήσουμε προς την Ολομέλεια ε, διότι διαφορετικά γελιοποιούμε το Κοινοβούλιο αν δεν μπορούμε να λάβουμε μία απάντηση ή μία απόφαση. Η κυρία κυρια να φέρθει και στην εμπορική θέση του Ισραήλ και πιστεύω ότι αυτό το θέμα μπορεί ε, να ε, επιληθεί με διάφορους τρόπους που προτείνει η νομική υπηρεσία και βεβαίως θα πρέπει η συμφωνία να επεκταθεί και στα εδάφη του Ισραήλ τα οποία αναγνωρίζουμε σύμφωνα με ε, την διεθνή νομοθεσία και όπου μπορεί να ισχύσει νομότυπα. Ε, ε, πιστεύω ότι υπάρχει ολιγορία, οι λόγοι είναι σαφείς, η κατάσταση στη Μέση Ανατολή είναι πάρα πολύ περίπλοκο για να επιλέξουμε εμείς ποιοι είναι οι καλοί και ποιοι οι κακοί και το να λέμε ότι το Ισραήλ ευθύνεται αποκλειστικά για την αποτυχία του, της ειρηνευτικής συμφωνίας ναι φέρει ευθύνες αλλά όχι αποκλειστικά ε, και ε, ε, υπερψηφίσαμε τη συμφωνία για την εμπορική συμφωνία με την Παλαιστίνη δεν βλέπω γιατί να καθυστερήσουμε λοιπόν και πιστεύω ότι το ίδιο πρέπει να γίνει και με την έκθεση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου διότι διαφορετικά δεν μπορούμε να προχωρήσουμε στην ε, ψήφιση αυτής της συμφωνίας που πρέπει να προχωρήσει στην Ολομέλεια με κάθε τρόπο. Ο κύριος Κοστέλε, ο οποίος είναι υπεύθυνο, ε, ε, πρόεδρος της Επιτροπής των Σχέσεων με την Παλαιστίνη. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, δεν είμαι μέλος αυτής της Επιτροπής, αλλά θέλω να δράξω την ευκαιρία να συνεισφέρω και εγώ σε αυτή τη συζήτηση. Όπως υπόθηκε, έγινε κάποια συζήτηση εδώ σε σχέση με το αν το θέμα είναι νομικό ή πολιτικό και ενώ τα νομικά θέματα ε, ρυθμίζονται δυνάμει της γνωμοδότησης ε, που έχουμε ενώπιόν μα. συμφωνώ με την κυρία Ντεκάιζερ και την άποψή τη ότι είναι πολιτική απόφαση ε, την οποία αντιμετωπίζουμε την περασμένη εβδομάδα ε, στην Επιτροπή αυτή συναντηθήκαμε με τον Υπουργό Εξωτερικών της ε, Παλαιστίνης ο οποίος μας μίλησε για την πολιτική τελμάτωση εκεί για τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη και ακούσαμε ανθρώπους που μας ε, είπαν ε, εδώ ότι πρόκειται για τιμωρία του Ισραήλ. Όχι, δεν πρόκειται για τιμωρία του Ισραήλ, αλλά θέλουμε να στείλουμε ένα ισχυρό μήνυμα και ένα ισχυρό πολιτικό μήνυμα. Ε, εγώ από τότε που ήρθα στο Κοινοβούλιο πριν λίγες εβδομάδες είχαμε πολλές προτάσεις σε σχέση με τις περαβίες των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και κάναμε και ε, κάποιες ισχυρές δηλώσεις για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τίποτα δεν σημαίνουν όλα αυτά αν δεν τα ε, στηρίξουμε και με πράξεις και μάλιστα η συνδίκη της Λισαβόνας μας υποχρεώνει να το κάνουμε και εγώ θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ ισορροπημένη η έκθεση της κυρίας Δεκάιζερ και Νομίζω ότι ε, η πρόταση να έχουμε μια ενδιάμεση έκθεση μπορεί να αντιμετωπίσει το θέμα της διαδικασίας των επικισμών και της παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και νομίζω ότι είναι καλύτερη η οδός που θα μπορούσε να ακολουθηθεί στο στάδιο αυτό. Έτσι λοιπόν, βάσει όσων είπε η κυρία Ντεκάιζερ, εγώ θα υποστήριξα την ε, έκθεση της εισηγήτριας ε, και θα έλεγα ότι πρέπει να πάρουμε μια πολιτική απόφαση από αυτού. συνάδελφος Μπέλντερ και ολοκληρώνονται οι παρεμβάσεις των κυρίων βουλευτών εδώ. Eh, λοιπόν, συμφωνώ με αυτά τα οποία μόλις είπε η επικεφαλής της ε, αντιπροσωπείας για την Παλαιστίνη, δηλαδή να αποφασίσουμε και ε, εκεί πρέπει να προχωρήσουμε, πρέπει να κλείσουμε αυτό το φάκελο που ήδη εκρεμεί εδώ και δύο χρόνια και είναι πραγματική ε, ντροπή για το κοινοβούλιο αυτό ότι καθυστερούμε και ολιγορούμε και παρουσιάζουμε συνεχή επιχειρήματα αλλά τώρα ορίμασε το θέμα, το και από την κυρία Λάτφορτ είναι ένα πολύ περίπλοκο θέμα και γι' αυτό πιστεύω ότι ανάλογα πρέπει να αντιδράσουμε. Εμείς πάντως θέλουμε όσο γίνεται πιο γρήγορα να πάει το θέμα στις αρμόδιες επιτροπές. Ευχαριστώ. Λοιπόν, ευχαριστώ. Εγώ συνήθω όταν ε, ασκώ την Προεδρία δεν παίρνω το λόγο, αλλά ήθελα να κάνω μια τεχνική ερώτηση για να κατανοήσω καλύτερα τη βούληση της εισηγήτριας, της κυρίας Δεκάιζερ. Αυτή η αναβολή, αυτό το πάγωμα που ζητάτε εσείς, ε, θα γίνει βάσει κάποιων όρων, εξαρτάται από κάτι ή όχι. Και ε, αναφέρεστε στο χρόνο, σε μια προθεσμία δύο ετών. Είναι μια δεσμευτική η προθεσμία αυτή χρονικά ή όχι. Θα ήθελα να μας πείτε κάτι σχετικά με το θέμα. Ε, punto... Και σε αυτό το σημείο να ρωτήσω αν η Κομισιόν που εκπροσωπείται από τον Άρθρο Λόπιαν θα ήθελε το λόγο. Ευχαριστώ. Θα είμαι πολύ σύντομα. Σάλτο Λόπιαν ονομάζομαι από τη Γενική Διεύθυνση Εμπορίου. Διαπραγματευτήκαμε για την συμφωνία αυτή προστήριξη των επιχειρήσεων. Η ΙΑΚΑ έχει εγκριθεί από τις νομικές υπηρεσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, έχει εγκριθεί από τρεις νομικές υπηρεσίε και των τριών δηλαδή θεσμικών οργάνων, Συμβουλίου, Επιτροπή και Κοινοβουλίου. Για τι διαπραγματεύσει θέλω να σας πω ότι επιβεβαιώθηκε πως έγιναν οι διαπραγματεύσεις σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο και το Κοινοτικό Δίκαιο, οπότε το θέμα του να ανοίξουμε ή να τροποποιήσουμε ε, την συμφωνία είναι κάτι εντελώς θεωρητικό, δεν είναι προς το συμφέρον μας. Εμείς έχουμε αναλύσει το θέμα και την ανάλυση αυτή σας την έχουμε παρουσιάσει και εδώ. Το δεύτερο θέμα είναι το θέμα της εφαρμογής. Η νομική υπηρεσία είπε ότι όλα τα θέματα μπορούν να τεθούν στο θέμα της εφαρμογής βάσει μηχανισμών και λοιπά που προβλέπονται στην ε, συμφωνία. Οπότε δεν τίθεται τίποτα άλλο από τη δικιά μας την πλευρά. Εμείς πιστεύουμε ότι μπορεί να μπορείτε να συμφωνήσετε ως έχει με τη συμφωνία αυτή. Μάλιστα, η συγκήτρια παρακαλώ και πέντε λεπτά για να απαντήσει. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν θα απαντήσω βέβαια σε όλες τις ερωτήσεις. Θέλω όμως να διευκρινίσω κάποια σημεία που άκουσα. Πρώτον, κατά πόσο εδώ τιμωρούμε το Ισραήλ. Όχι, δεν πρόκειται περί αυτού, δεν πρόκειται για μια τιμωρία, για μια κύρωση. Απλώς τοποθετούμεθα σε σχέση με ένα de facto upgrading, μια αναβάθμιση που γίνεται de facto, δεδομένου ότι δίνουμε νέες δυνατότητες στο Ισραήλ. Στη νέα πολιτική γυτνίασης. Η ιδέα είναι να βάζουμε προϋποθέσεις σε σχέση με την πρόθεση παρετέρω στοιχείων στα πλαίσια μιας συμφωνίας που έχουμε ανάλογα με το τι θέλουμε να πετύχουμε. Από το Ισραήλ προς το παρόν δεν μπορούμε να πετύχουμε την ειρήνη, γιατί η ειρήνη δεν εξαρτάται μόνο από το Ισραήλ. Όμως, οι επικισμοί, ναι, εξαρτώνται από το Ισραήλ. Οι κυβερνήσεις του Ισραήλ, κάποιες περισσότερο από άλλες, ευνόησαν τους επικισμούς. Δεν έχουν να κάνουν επικισμοί με το αν οι διαπραγματεύσεις θα συνεχιστούν ή όχι και το ε, μπλοκάρισμα της Γάζα δεν εξαρτάται από αυτό. Τα προϊόντα που λέμε ότι πρέπει να απαγορεύονται έχουν να κάνουν μόνο με το Ισραήλ. Συνεπώς, όταν ορισμένοι έρχονται και μου λένε «Μα δεν μπορείτε να τιμωρείτε το Ισραήλ για την ειρήνη που δεν υπάρχει», συμφωνώ απόλυτα με αυτό. Αλλά όταν μου λένε «Δεν μπορείτε να ζητήσετε από το Ισραήλ μια ατζέντα για τα ανθρώπινα δικαιώματα για να δώσουμε κι εμείς κάτι, με αυτό δεν συμφωνώ. Η νέα πολιτική γυτνία τι είναι για ορισμένους και όχι για άλλους. Μου λένε για το Ισραήλ δεν πρόκειται να λειτουργήσει γιατί δεν θα αλλάξει τίποτα. Ε, άμα δεν αλλάξει τίποτα, τότε έχουμε σοβαρό πρόβλημα με το Ισραήλ. Αν το Ισραήλ μπορεί να θέλει να μην αλλάξει τίποτα όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, ενώ από άλλε χώρε αυτό το ζητάμε, ε, τότε λέω έχουμε πρόβλημα με το Ισραήλ. Και δεν μιλάω με τη δυσκολία του να αρχίσουν και πάλι οι ειρηνευτικέ διαπραγματεύσει. Συνεπώ, το να λέμε ότι δεν θα πάρουμε τίποτα από το Ισραήλ όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι σκανδαλώδε. Και το λέω εδώ ξεκάθαρα. Και γι' αυτό δεν καταλαβαίνω. Εδώ στο Κοινοβούλιο, στην Επιτροπή μας και όπως μας το γνωστοποίησε και το ΕΛΚΑ θα υπάρξουν ψηφοφορίε για τη διαπραγμάτευση των συμφωνιών από την άλλη θα υπάρξουν και τροπολογίες που θα είναι κατά τη συμφωνίας αυτής, ακριβώς επειδή είναι αδύνατο να πετύχουμε κάτι από το Ισραήλ ε, για τα θέματα στα οποία αναφέρονται στη συμφωνία σύνδεσή μας και που δεν έχει να κάνει με τις ειρνευτικές διαπραγματεύσεις. Τώρα για τα τεχνικά και νομικά ζητήματα. Διάβασα την ε, νομική γνωμοδότηση ξανά και ξανά Εννοείται, μπορούμε να συνεχίσουμε σαν να μην τρέχει τίποτα. Δηλαδή, το Ισραήλ λέει, α, είναι τα δικά μου εδάφη και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει να κάνει ό,τι έκανε πάντα, δηλαδή να λέει ναι, αλλά όχι, για μας δεν είναι κτλ. Το θέμα όμως της εφαρμοσιμότητας, τι αποτέλεσμα έχει επιτόπου. Μηδέν στο πηλίκον. Τα προϊόντα των επίκων τελικά πάντα θα μας έρχονται. Ό,τι δηλαδή κάναμε μέχρι τώρα δεν έχει αποφέρει καρπούς. Και γι' αυτό λέμε ότι για να έχουμε μια θέση αναδίπλωση συμβιβαστική, γι' αυτό ακριβώς και εγώ στο σχέδιό μου, σχέδιο γνωμοδότησης, περιλαμβάνω κάτι πιο τεχνικό χαρακτήρα. Δηλαδή είναι αυτή η προσωρινή έκθεση. Τι είναι όχι, δεν είναι αναβολή και τα λοιπά τη συμφωνίας. Όχι. Αν αποφασίσετε ότι το... δεν μας ενδιαφέρει το πολιτικό μήνυμα και τη θέλουμε τη συμφωνία, ε, θα την έχετε αυτή τη συμφωνία. Αλλά τότε αυτό που θέλω είναι επιτόπου να αλλάξουν τα πράγματα όσον αφορά τα εζελινά προϊόντα. Και γι' αυτό και αυτή η ενδιάμεση έκθεση, η οποία είναι μια έκθεση που πρέπει να κάνει ίντα, όχι εμείς. Υπάρχει το άρθρο 81 του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε σχέση με αυτά, ο οποίος λέει ότι η προσωρινή έκθεση χρησιμεύει για να συμπεριλάβει συστάσεις όσον αφορά την τροποποίηση ή την εφαρμογή της προτινόμενης πράξης. Δηλαδή μια προσωρινή έκθεση χρησιμεύει είτε για να επαληθεύσει την εφαρμογή είτε για να προτείνει μια τροποποίηση. Η τροποποίηση που σας πρότεινα πριν, στην περίπτωση που κερδίσει το ναι, για παράδειγμα θα ήταν να εισάγουμε ευθύ εξ αρχή, χωρί να επαναπραγματευτούμε όλη την ε, έκθεση, αυτή τη μικρή πρόταση. Εάν εσείς αποφασίσετε, παρόλα όσα έχουν ακουστεί εδώ, αν αποφασίσετε να περάσει η συμφωνία αυτή, δεν θα ήθελα επιπλέον να μπούμε σε δυσκολία όχι νομιμότητα τυπικά, αλλά να εθελοτυφλούμε, γιατί σήμερα δεν έχουμε κανέναν τρόπο για να ελέγξουμε την εισαγωγή προϊόντων από τους επικισμούς στην Ευρώπη. Και δεν θα μας ε, βοηθήσουν δηλώσεις που λένε όχι εμείς δεν αναγνωρίζουμε τους επικισμούς που θα αλλάξει και κάτι. Όχι, κάτι πρέπει να αλλάξει στη συμφωνία. Και εγώ σας έδωσα έναν τρόπο για να το κάνουμε αυτό, για το οποίο με σε και κάποιο νομικό. Θα μπορούσε να βοηθήσει. Αλλά έτσι κι την έκθεση αυτή θα πρέπει να την κάνει ίντα και όχι εμεί. Είναι μια θέση αναδίπλωση. Σα την προτείνω. Πιστεύω ότι δεν θα μπορέσουμε να έχουμε πολιτικό συμβιβασμό. Μπορούμε στα τεχνικά στοιχεία να πετύχουμε συμβιβασμό, αλλά εδώ πολιτικό συμβιβασμό δεν πιστεύω ότι θα πετύχουμε για την συμφωνία αυτή. Αυτά είναι τα συμπεράσματά μου. Συνεπώς, ε, πρόεδρε, συγγνώμη, η ερώτησή σας ποια ακριβώς ήταν, γιατί εγώ ήθελα να απαντήσω. Αν ε, το έτοιμά σας ε, για πάγωμα, για αναστολή, αν κατά κάποιο τρόπο συνδέεται με κάποιες συγκεκριμένες προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται και αν η προθεσμία των δύο ετών είναι μια προθεσμία, ένας προθεσμία οριστή, να το προτείνεται για κάποιο λόγο. Euh, Πρόεδρε, δεν πρότεινα ούτε πάγωμα, ούτε δύο έτη. Η Ίντα το προτείνει αυτό, όχι εγώ. Εγώ πρότεινα, ανακοίνωσα τροπολογίες και πρότεινα και μία λύση αναδίπλωσης, η οποία ζητάει να εκπονηθεί μία ενδιάμεση έκθεση. Και σας το είπα προφορικά, γιατί δεν μπορώ να σας το πω γραπτά, ότι θα μπορούσε να περιλαμβάνει μια ελάχιστη τροποποίηση η οποία δεν απαιτεί αναθεώρηση ολόκληρης της συμφωνίας. Δεν πρότεινα πάγωμα. Είπα ότι είναι καλύτερα να μην το εξετάσουμε αυτό το θέμα αυτή την εποχή. Οι πολιτικές ομάδες όμως αποφάσισαν κάτι διαφορετικό. Συμμορφώνομαι, αλλά δεν προτείνω πάγωμα και δεν προτείνω προϋποθέσεις. Δεν έχω την πολιτική δυνατότητα να βάλω προϋποθέσεις και όρους. Λέω όμως ότι μία προσωρινή έκθεση δεν παγώνει απολύτως τίποτα και αφορά μία ή μικρή τροποποίηση ή διευκρίνηση εφαρμογής. Από εκεί και πέρα η ίντα θα αποφασίσει για το τι θα κάνει. Προθεσμία για τις τροπολογίες 29 Μαρτίου 12 το μεσημέρι. Και να περάσουμε τώρα στο σημείο 4, η χρήση των δεδομένων που περιέχονται επιβατών. Έχουμε τη συντάκτη της νομοδότησης, είναι η κυρία Λάτφορτ. Η συγκίτρια έχει προετοιμάσει ένα σχέδιο γνωμοδότησης. Όποιος ε, δεν ενδιαφέρεται να απομακρυνθεί παρακαλώ, αλλά με ησυχία. Λοιπόν, η συγκέντρια επικεντρώθηκε στις τροπολογίες που προτείνονται μόνο στις πτυχές που αφορούν απευθείας τις αρμοδιότητες της Επιτροπής μας. Ο στόχος ε, είναι να συνεισφέρει στην αρμόδια Επιτροπή, όχι να υπάρχει επικάλυψη του έργου της Επιτροπής. Σας παρακαλώ, μπορείτε να δώσετε λίγη προσοχή και να σεβαστείτε και ποιον παραμένει και θέλει να εργαστεί η ανταλλαγή απόψεων στην Επιτροπή μας ε, θα γίνει σήμερα, άπαξ. Και θα δώσω τώρα το λόγο στην ε, Βαρόνι Λάτφορτ. Παρακαλώ. Μικρόφωνο παρακαλούμε. Όπως σωστά είπατε, Πρόεδρε, όπως ε, είπατε πολύ σωστά κύριε Πρόεδρε, ε, πρέπει να εξετάσουμε τις ε, εξωτερικές επιπτώσεις την, της οδηγίας του συστήματος PNR. Όχι δηλαδή η συμφωνία του Αμερικανικού PNR που, που ψηφίσαμε σήμερα το πρωί στην Επιτροπή Ελευθεριών. Οπότε κοίταξα να δω ποιες είναι οι εξωτερικές πτυχές οι οποίες πρέπει να τονιστούν. Βεβαίως ε, το πλαίσιο είναι ότι υπάρχουν πολλά ψηφίσματα και ε, ανέρχονται σε μία δεκαετία. Έχουμε τονίσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την ανάγκη να υπάρξει μία συλλογή των στοιχείων PNR ε, σε ένα πλαίσιο και ε, να συσχετιστούν με τα ανθρώπινα δικαιώματα των πολιτών και να εξασφαλίσουμε ότι τα στοιχεία αυτά θα χρησιμοποιούνται μόνο για λόγους εφαρμογής ε, της, ε, του νόμου και δεν θα χρησιμοποιούνται για εγκληματικούς σκοπούς. Επίσης, Υπάρχουν συμφωνίες με τρίτες χώρες οι οποίες πρέπει να συνάδουν με τις δικές μας προδιαγραφές. Παρακαλώ όσους ε, είναι όρθιοι στην αίθουσα και μιλούν να εγκαταλείψουν την αίθουσα γιατί ε, δεν μας βοηθούν. Άρα, ο στόχος αυτής της οδηγίας ε, είναι ε, να προχωρήσει στην Επιτροπή Ελευθεριών όπου ο συνάδελφός μου και συμπατριώτης μου κύριος Κιάρκοπ είναι εισηγητής και ε, ένας από τους λόγους για τους οποίους ζήτησα να συντάξω μία γνωμοδότηση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων αναφέρεται στις σχέσεις των διαφόρων αεροπορικών εταιριών με τις ε, ε, χώρες της σημαίας του κάθε αερομεταφορέα και είπα ότι στο τέλος της μεταβατικής περίοδου όταν δηλαδή έπρεπε τα στοιχεία αυτά να προωθηθούν προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, εάν υπάρχουν τεχνικά προβλήματα να αντιμετωπιστούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να προσπαθήσουμε να αποφύγουμε με μονομένες πρωτοβουλίες των κρατών μελών. Θέλω δηλαδή να εξασφαλίσω ότι θα υπάρχει μία προσέγγιση κοινοτική προς τις συναλλαγές με τις αεροπορικές εταιρείες. Δηλαδή δεν θέλουμε να έχουμε διαφορετικές αντιμετωπίσεις από τα διαφορετικά κράτη-μέλη. Και στην ε, τροπολογία 2 τόνισα το ότι τα δικαιώματα των επιβατών θα πρέπει να εφαρμόζονται και στους πολίτες Ευρωπαϊκής Ενώσεως και σε αυτούς των τρίτων χωρών ή δηλαδή σε οποιοδήποτε επιβάτη βρίσκεται μέσα στην επικράτεια ασχέτως της υπηκότητας του. Ε, υπηκότητάς του. Στην τροπολογία 3 τονίζω ότι δεν συμφωνώ με την συμπερίληψη των εσωτερικών πτήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό το λέω από την αρχή. Ο στόχος αυτός θα εξεταστεί ως προς την ουσία στα πλαίσια της συζητήσεως στην Επιτροπή Ελευθεριών αλλά είπαμε ότι αναφερόμαστε στις σχέσεις του αερομεταφορέα με το κράτος της σημαίας και ε, θέλουμε να έχουμε εφικτές μεταβατικές διατάξεις και να μπορέσουμε να μην ε, επιβαρύνουμε υπερβολικά την εφαρμογή που θα δυναμητήσει την εφαρμογή του συστήματος PNR. Οπότε θέλω να συζητήσω με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να προσπαθήσουμε να κάνουμε τα πρώτα αργά βήματα προτού αρχίσουμε ε, να ε, επιταχύνουμε να αφήσουμε δηλαδή ορισμένα θέματα προς επίλυση σε μία μετέπειτα χρονική στιγμή όσον αφορά την τροπολογία 482 λέω ότι η Διεθνή Συμφωνία πρέπει να προσφέρει εχέγγυα που θα συνάδουν με αυτήν την οδηγία και αυτό προσπαθήσαμε να κάνουμε και μέχρι στιγμής στη συμφωνία. Ε, ξέρω ότι υπάρχει αυτό το θέμα. Έχω και εγώ ανησυχίες ε, διότι υπερψήφισα σήμερα το πρωί στην Επιτροπή Ελευθεριών ορισμένα από αυτά τα θέματα ε, εις βάρος των εναλλακτικών λύσεων. Οι συμφωνίες δεν είναι ακριβώς το ίδιο με την, την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία αλλά πρέπει να μπορούν να είναι συνεκτικές και γι' αυτό στην τροπολογία 6 ζητώ να επεκτείνουμε τον αριθμό πληροφοριών που μας παρουσιάζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με την εφαρμογή από τους αερομεταφορείς τρίτων χωρών της συμφωνίας και σχετικά με τη μεταβίβαση των στοιχείων σε τρίτες χώρες για να εξετάσουμε ε, πόσο συχνά υπάρχουν ε, τέτοιες ε, μεταφορές και πέραν αυτού είμαι στη διάθεσή σας για να απαντήσω σε οποιαδήποτε ερώτηση. Ευχαριστώ. Συνάδελφος Φαγιάν, δύο λεπτά η κυρία Φαγιάν. Ευχαριστώ. Καταρχήν, θέλω να ευχαριστήσω τη συνάδελφο Σάρα, που στηρίζω τις περισσότερες από τις θέσεις της, στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ. Ασχολούμαστε με όλα αυτά τα θέματα και πιστεύω ότι ο στόχος ε, της προτινόμενης ε, οδηγίας είναι η καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Έχουμε δυνατότητα για ένα συντονισμένο σύστημα, αλλά υπάρχει μια σειρά αμφιβολιών, υπάρχουν αποκλίνουσες απόψεις, χρειαζόμαστε ανάλυση των δεδομένων, χρειαζόμαστε ονόματα, διευθύνσεις, τραπεζικά δεδομένα, αριθμούς διαβατηρίων κτλ. Συμφωνώ ότι πρέπει να είμαστε αποφασιστικοί στην ε, ε, καταπολέμηση της τρομοκρατίας, αλλά θα πρέπει να διασφαλίσουμε και την προστασία των δεδομένων. Πρέπει να προστατεύσουμε αυτά τα προσωπικά δεδομένα προκειμένου να αποφύγουμε την παραβίαση των δικαιωμάτων Και επίσης πρέπει να έχουμε μία ολοκληρωμένη προσέγγιση για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Αυτά τα δεδομένα πρέπει να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και την καταπολέμηση της τρομοκρατίας ε, και όχι για άλλα εγκλήματα. Αυτό ήταν ένα από τα μεγάλα προβλήματα στην ε, περίπτωση της σύναυσης της συμφωνίας με τις ΕΙΠΑ που υποστηρίχθηκε σήμερα. Σε ό,τι αφορά τώρα το κόστος, θα ήθελα να προσθέσω ότι υπάρχουν ε, πολλές αμφιβολίες σχετικά με το κόστος, ανεξάρτητα με το αν θα γίνεται επεξεργασία των δεδομένων για τις εξωτερικές πτήσεις. Ό,τι αφορά τις εξωτερικές πτήσεις δεν έχει κανένα νόημα. Το κόστος θα ήταν πάρα πολύ υψηλό για τις μικρότερες χώρες, πιστεύω ότι χρειαζόμαστε ένα κεντρικό σύστημα, αλλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει αγγίξει καθόλου το θέμα αυτό. Και υπάρχει και κάτι άλλο, στο οποίο θέλω να επιστήσω την προσοχή σας. Στην τελευταία μελέτη της ε, Ένωσης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, η μελέτη αυτή επικρίνει αυτή την προτενωμένη οδηγία, ζητήσαμε και την γνωμοδότηση σε άλλους συναδέλφων ε, στη ΛΕΙΜΠΕ, αλλά ε, υπάρχει ε, κάποια απόκληση απόψεων και χρειαζόταν περισσότερο χρόνο. Μάλιστα, κυρία Λόπες, δύο λεπτά μόνο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αυτό το εργαλείο, αυτό το μητρό, ε, ουσιαστικά ακολουθεί ε, το μητρό τη συμφωνία που υπογράψαμε σήμερα με τον Ήπειρο. Πρόκειται για ένα μέσο καταπολέμηση ε, του εγκλήματο, αλλά πραγματικά αντίκειται στα συντάγματα των 27 κρατών μελών και στη συνθήκη τη Λισαβόνα. Γιατί εκεί υπάρχει η προστασία, προβλέπεται η προστασία ενώ προσωπικών δεδομένων ο Ευρωπαίος Επόπτης ε, για το άρθρο 29 της ε, πρώην οδηγία προστασία ε, των Δεδομένων επέκρινε τη μορφή αυτού του Μητρώου. Δεν επιτρέπονται όλα για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Το σύστημα που αναλύει τη συμπεριφορά των πολιτών μας μετατρέπει όλου σε Είναι ορολογιακή βόμβα κατά του κράτου δικαίου. Εγώ θυμάμαι τι είπε ο ποινικό. Λόγος Μπεκαρία ότι είπε ε, καλύτερα να είναι ένας ένοχος στο δρόμο παρά ένας αθώος στη φυλακή. Μόνο το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία έχουν βάλει αυτό το σύστημα ε, στο νομοθετικό τους σύστημα κατά των μεταναστών. Μόνο με καταπολέμηση της τρομοκρατίας πρέπει να γίνεται ε, μόνο σε πολύ συγκεκριμένες περιόδους θα πρέπει να εφαρμόζεται αυτό το σύστημα όμως η δικαστική παρέμβαση είναι απαραίτητη για να είμαστε σίγουροι ότι γίνονται σεβαστά τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κόστο δεν είναι ένα θέμα που πρέπει να δούμε εδώ. Αν πράγματι πρόκειται για μια διαδικασία που είναι απαραίτητη, σίγουρα τα κράτη-μέλη θα θέσουν και την απαραίτητη χρηματοδότηση. Α ξεκινήσουμε με την τρομοκρατία και ίσω ε, θα καταλήξουμε εκεί, γιατί δεν πρέπει να καταστρέψει το κράτο δικαίου μα ε, ο αγώνα κατά τη τρομοκρατία, κατά του εγκλήματο. Ευχαριστώ δεν ε, θα έλεγαν ε, μια παράθεση του Μπακαρία πολύ Ιταλή. Παρακαλώ, συνάδελφος Ντάρμουτ. Microphone. Microphone. Uh, no. No. Here's another one. Here's the next one. The, uh, the uh, ο Earl of Dartmouth. Ε, πρέπει να σας πω ότι μπορούμε να συνοψίσουμε το στόχο η στην εισαγωγή, διότι ο στόχος είναι η καταπολέμηση της τρομοκρατίας, αλλά και η προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και συνοψίζει τη θέση άλλης επιτροπής λέγοντας ότι η μετάδοση των στοιχείων PNR θα περιοριστεί στις απαραίτητες περιπτώσεις ε, για πολύ σοβαρά αδικήματα και αυτό το αντιπαραθέτω με το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης όπου και στις δύο περιπτώσεις υπάρχει μετάδοση ε, ε, δεδομένων και σε αντίθεση με το Ευρωπαϊκό Ένταλμα εδώ δεν υπάρχει κανένα αχέντιο και υπάρχουν άτομα και ακόμη και Βρετανοί πολίτες μπορούν να μεταφερθούν σε φυλακές αμφιλεγόμενες σε πολύ απεχθή συστήματα πολιτικά και δεν υπάρχει καμία εγγύηση η οποία υπάρχει στο ευρωπαϊκό στο Ευρωπαϊκό Ένταλμα Οπότε βλέπετε εδώ τη διαφορά. Σύμφωνα με τη Βαρόνη Λάτφορτ και τους συνεργάτες της υπάρχει ε, ένα ε, αίσθημα αγαλιάσεω διότι μπορέσατε να περιορίσετε την πρόσβαση ε, στα ευρωπαϊκά δεδομένα. Αλλά τι είναι πιο βασικό, οι άνθρωποι ή τα δεδομένα. Διότι όσο προχωρούμε περισσότερο προς ένα υπερκράτος ευρωπαϊκό τόσο μειώνουμε την αξία του πολίτη. Αυτά είχα να σας πω. Κύριε Αυλάκη, πολύ σύντομα. λεπτό. Έχω μία ανησυχία σχετικά με την πρόταση αυτή και ελπίζω το Κοινοβουλίο να την απορρίψει ή να την διορθώσει επί της ουσίας. Οι συνάδελφοι ήδη τοποθετήθηκαν ε, σχετικά με την ομιμότητα αυτού του μέσου, αλλά θα έλεγα ε, απλώς ε, κάτι για την πλήρη χρησιμοποίηση του στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Εγώ ως εμπειρογνώμονας για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος της τρομοκρατίας δεν πιστεύω ότι είναι το κατάλληλο μέσο αυτό. Εδώ διακινδυνεύουμε να ακολουθήσουμε την αμερικανική παράνοια. Συγγνώμη, υπάρχει μία ε, βοή εδώ από κάτω και μοιάζουμε περισσότερο όχι με κοινοβούλιο αλλά με δισκοτέκ. Δηλαδή ακούγεται μία μουσική. Να τη σβήσουμε αυτή τη μουσική. Να κλείσουμε τις πόρτες. No, posso invitarvi a Μπορούμε να κλείσουμε τις πόρτες. Σας παρακαλώ. Πρέγω. Αρλάκη. Yes, I was... Κύριε Αρλάκη. Ναι, έλεγα ότι φοβάμαι πως ακολουθούμε εδώ την Αμερικανική στρατηγική και φιλοσοφία για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του οργανού που ουσιαστικά εκείται στο να δημιουργούνται αυτές οι τεράστιες βάσεις δεδομένων που ποτέ δεν απέδειξαν την ε, αποτελεσματικότητά τους. Ε, οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις και αρχές επιβολής ε, του νόμου από την 11η Σεπτεμβρίου ακολούθησαν διαφορετική στρατηγική. Δηλαδή χρησιμοποιούσαν επιλεκτικά δεδομένα, τις μυστικές πληροφορίες, τις έρευνες. Ποτέ δεν χρησιμοποίησαν αυτές τις τεράστιες βάσεις δεδομένων γιατί η χρησιμότητά τους είναι κάτι αμφισβητήσιμο και έχει φανεί ότι ούτε ένας μαφιόζος, ούτε ένας τρομοκράτη, δεν έχει συλληφθεί ε, βάσει αυτών των μέσων. Οι διοκτικές αρχές αυτή την Ήπειρο ήδη έχουν στη διάθεσή τους όλα τα στοιχεία που θέλουν σε, ε, για τους ύποπτους ανθρώπους ε, και ξέρουν τι κάνουν οι άνθρωποι αυτοί. Δεν χρειάζεται να αυξήσουμε σε καμία περίπτωση τον αριθμό των ε, παραβιάσεων, ε, ούτε πρέπει να ακολουθήσουμε αυτή την κατεύθυνση παραβιάζοντα την ελευθερία. Της ελευθερίας ευχαριστώ. Κύριο Σουνγκουρεάνου. Ένα μισή λεπτό, σας παρακαλώ, και να δώσουμε το λόγο και στον κύριο Λούνατσεκ μετά. Ευχαριστώ. Συμφωνώ με όσα υπόθηκαν. Ε, από την συγκήτρια εκτός από την τροπολογία 5 ότι τα κράτη-μέλη μπορούν να διαβιβάζουν τα δεδομένα PNR σε μια τρίτη χώρα μόνο αν ε, έχει γίνει μια έρευνα στη χώρα αυτή. Ε, υπάρχει ένας περιορισμός που σημαίνει ότι τα δεδομένα PNR θα διαβιβάζονται μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Αυστραλία και νομίζω ότι θα ήταν πιο σοφό να χρησιμοποιήσουμε κανόνες που θα επιτρέπουν την αλλαγή των δεδομένων ε, PR ε, ανά περίπτωση. Φυσικά αυτό δεν ε, πρέπει να σημαίνει ότι η διαβίβαση των δεδομένων θα επιτρέπεται απαραίτητο. Θα πρέπει να επιτρέπεται να γίνεται στις χώρες αυτές που διασφαλίζουν την επαρκή προστασία των δεδομένων και φυσικά με την συνένεση του κράτου μέλους από το οποίο αποκτήθηκαν τα δεδομένα αυτά. Ευχαριστώ. Πολύ ωραία. Λούνατσα και μισή λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εν ονόματι τη ομάδα μου θα ήθελα να σα πω από την αρχή ότι η ομάδα μου έχει τι ίδιε δυσκολίε με τον κύριο Αλάκινε σχετικά με την ανάγκη και την αναλογικότητα τη συλλογή αυτών των δεδομένων όπου αναφέρονται στου επιβάτε. και ιδίω σε σχέση με αυτό που προτείνει σαν τροπολογίε η κυρία Λάτφορτ λίγε από αυτέ μα βρίσκουν σύμφωνου όσον αφορά την προστασία των δεδομένων διότι δεν πρέπει να καλύπτονται μόνο οι πολίτες Ευρωπαϊκής Ενώσεως αλλά και τρίτων χωρών. Το πρόβλημα μου όμως σχετικά με την πρόταση αυτή γενικώ είναι ότι για τη δικιά μου πολιτική ομάδα δεν είναι προφανές δεν θέλουμε όλα αυτά τα στοιχεία για να καταποτελήσουμε την τρομοκρατία και ακόμη και αν οι τρίτες χώρες αυτές έχουν συμφωνίες μαζί μας είτε πρόκειται για την Αυστραλία είτε για τον Καναδά αλλά με τους άλλους ποιος μπορεί να ελέγξει ότι υπάρχει σωστή εφαρμογή της συμφωνίας δεν φτάνει να υπογραφεί η συμφωνία. Πρέπει να υπάρχει προστασία δεδομένων των πολιτών που είναι εξίσου σημαντική όσο η καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Η στήριξή μας λοιπόν βαίνει προς την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, όχι όμως στη χρησιμοποίηση της μέθοδου αυτής για να πατάξει κανείς την αντιπολίτευση σε ορισμένες χώρες. Γι' αυτό και η πολιτική η ομάδα έχει πολλές επιφυλάξεις και στα πλαίσια αυτά θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε σχετικά με τις τροπολογίες, αλλά αυτή τη στιγμή δεν είναι κάτι το οποίο μπορούμε να δεχθούμε γενικώ. Ευχαριστώ. Σας υπενθυμίζω ότι η προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών είναι στις 21 του μήνα. Λοιπόν, να περάσουμε στο επόμενο θέμα, ανταλλαγή απόψεων σε σχέση με τα εξωτερικά χρηματοδοτικά μέσα. Παρακαλώ, σας δω συγγνώμη. Ναι, με συγχωρείτε για να απαντήσετε, αλλά σας παρακαλώ, επειδή έχουμε καθυστερήσει, να είστε σύντομοι, γιατί εδώ και 20 λεπτά μας περιμένουν οι καλεσμένοι μας. Ναι, βεβαίως. Το κύριο θέμα για την αναγκαιότητα και την αναλογικότητα είναι κάτι που προσπαθώ να σας ξεκαθαρίσω ότι το θέμα αυτό εγώ δεν το αντιμετωπίζω παρά ως γνωμοδότηση της ΑΦΕΤ. Η επί της συζήτηση γίνεται στην ΛΥΜΠΕ έτσι κι αλλιώς. Οπότε διαφορετική είναι η δικιά μας η γνωμοδότηση. Έτσι κι αλλιώς Έχω συζητήσει ξανά και ξανά τις προτεραιότητες για το PNR και έχω ασχοληθεί και πριν από τρία χρόνια με το profiling της κατατομές που προτείνονται. Και εγώ θέλω τις δοκιμές αναγκαιότητας και αναλογικότητας, αλλά είναι θέμα πολύ περισσότερο της Επιτροπής Ελευθεριών του Πολίτη. το θέμα το πολιτικό, είτε πρόκειται για τους ελεύθερους στον Βασίλιο Βασίλειο, είτε πρόκειται για άλλα δεν είναι της παρούσης. Ελπίζω πάντως να ξέρουν και όσοι αναφέρθηκαν στο Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης τόσα όσα και εγώ. Τώρα αναφέρθηκε επίσης το κόστος. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, πάντα μας ΕΝΑΡ. Γιατί πάντα λέμε, ωραία, να συλλέγονται τα δεδομένα, Ποιο θα πληρώσει όμως γι' αυτά. Και οι αεροπορικές εταιρείε δεν θέλουν βέβαια να, βάλουν να αναλάβουν αυτές το κόστος και αυτό είναι θέμα όμως <clears throat> της ΛΥΜΠΕ. Για την κυρία Ρομερολόπε. Αναφέρθηκε στην αιτιολόγηση. Θα ξέρω όμω και εκείνη από την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ ότι τον όρο unknown suspect που χρησιμοποιεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η άγνωστη ύποπτη, ε, τη ζητήσαμε να το αλλάξουν. Τι θα πει αυτό άγνωστη ύποπτη, που είσαι ύποπτος και σε ξέρουν ή που είσαι άγνωστος. Θέλουμε να περιοριστούμε στην τρομοκρατία και τα σοβαρά εγκλήματα. Ο δικός μου δισταγμός πριν υπερψηφίσω τη συμφωνία με τις ΗΠΑ ήταν ότι πιστεύω ότι ερμηνεύονται διαφορετικά οι διάφορες ρήτρε της συμφωνίας. Και το είπα και την προηγούμενη εβδομάδα στην Ουάσιγκτον. Το θέμα του ελέγχου της εφαρμογής της συμφωνίας αυτής θα είναι ζωτική σημασία. Εγώ δεν νομίζω ότι οι ΗΠΑ και η Ευρώπη βρισκόμαστε στην ίδια συχνότητα όσον αφορά την ερμηνεία της συμφωνίας. Για την τροπολογία 5, ο κύριος Σουγκουριάνο μίλησε για αυτή. Εγώ δεν λέω ότι έχουμε συμφωνία με τις τρίτες χώρες. Οι άλλοι εναλλακτικοί είναι οι χώρες αυτές να πρέπει να, έχουν, να είναι συμβαλόμενα μέρη μιας διεθνούς συμφωνίας. Πάντως, αν υπάρχει κάτι ακόμα το οποίο δεν κάλυψε, ευχαρίστως διμερός να το καλύψω. Ευχαριστώ. Λοιπόν, ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τα εξωτερικά χρηματοδοτικά μέσα 2014-2020. Να καλωσορίσουμε και σα δώσω συγγνώμη για την καθυστέρηση. Να καλωσορίσουμε του καλεσμένου μα λοιπόν. Οι ομιλητές ε, που έχουμε προκαλέσει είναι η κυρία Μαρία Μερνάκη, διευθύνουσα Σύμβουλο Παγκοσμίων και Πολυμερών Θεμάτων τη Υπηρεσία Εξωτερική Δράση, ο κ. Στεφανό Σανίνο, Γενικό Διευθυντή για τη Διεύρυνση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο κ. Κλάου Ρουντισάουσερ. Συγγνώμη για την πώ προφέρω το όνομά ε, Διευθυντή για την Ποιότητα και τον Αντίκτυπο στην και του Τουν Κλάι Μάρκ, Διευθυντή της Υπηρεσίας για τα Μέσα άσκηση Εξωτερικής Πολιτικής της Κομισιόν. Αυτή είναι η πρώτη ανταλλαγή απόψεων για το νέο πακέτο εξωτερικών χρηματοδοτικών μέσων δηλαδή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το πακέτο υιοθετήθηκε στις 7 Δεκεμβρίου του 2011 και είναι σημαντικό αυτό το θέμα γιατί τα νέα χρηματοδοτικά μέσα ε, θα σηματοδοτήσουν ε, την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με την εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2014-2020. Αυτό αποτελεί ένα πακέτο προκειμένου να υπάρχει με καλύτερη συνέπεια, αποτελεσματικότητα και προβολή της θέσης του Κοινοβουλίου στο θέμα αυτό. Εγώ θα έλεγα να ξεκινήσουμε τη συζήτηση ζητώντα από την ε, εκπρόσωπο τη Υπηρεσία Εξωτερική Δράση να μα εξηγήσει ποια νέα θέματα έχουν εισαχθεί με τι προτάσει των νέων χρηματοδοτικών μέσων και ποιε είναι οι διαφορέ σε σχέση με τα σημερινά χρηματοδοτικά μέσα. Έτσι λοιπόν θα ήθελα να μας το ορισμένα οριζόντια στοιχεία όπως καταρχήν με ποιους όρους στις προτάσεις διευρύνεται ο ρόλος ελέγχου του Κοινοβουλίου των ε, χρηματοδοτικών μέσων για την εξωτερική δράση και ιδίως των ε, στρατηγικών αποφάσεων που συνδέονται με τα μέσα. Δεύτερον, κατά κάποιο τρόπο οι προτάσεις της Κομισιόν προωθούν τις αρχές της δημοκρατίας, του σεβασμού των ανθρώπινων δικαιωμάτων και ποιε είναι οι συμφωνίε συνεργασία μεταξύ τη Υπηρεσία Εξωτερική Δράση και τη Επιτροπή για τον προγραμματισμό και την εφαρμογή των μέσων αυτών. Τέταρτον, πώ ε, θα γίνει ο συντονισμό μεταξύ Ένωση και κρατών μελών και πώ θα ελοπιθεί ο συντονισμό μεταξύ των διεθνών οργανισμών και των διεθνών δωρητών ποιες είναι οι μορφές εταιρική σχέσης που έχουν προβλεφθεί με τις ε, χώρες δικαιούχους, ε, καθώς και πιθανή ευθυγράμμιση της Βοήθειας Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις πολιτικές προτεραιότητες και των ε, προγραμμάτων των χωρών προορισμού και με ποιους όρους οι μη κρατικοί φορείς και οι κοινωνία των πολιτών εμπλέκονται στην παρακολούθηση και στην εφαρμογή και ποια είναι η πρόοδος σήμερα και ποια πρόοδος προβλέπεται για το μέλλον. Λοιπόν, για να τα βάλουμε τη σειρά, θα δώσουμε κατόπιν το λόγο στους συντονιστές. Ε, τρία λεπτά στον καθένα. Συνάδελφοι Βιγγένιν, Κούκαν, Μπραντνερ και Μάουρο. Καταρχήν λοιπόν, από τους σοσιαλιστές, συνάδελφος Βιγκένιν για το μέσο πρωτεξιακής βοήθειας. Έχετε το λόγο. Thank you very much. Uh, Ευχαριστώ πολύ θα είμαι σύντομος, γιατί έχει περάσει ο χρόνος. Έχω όμως κάποιες παρατηρήσεις όσον αφορά το προταξιακό αυτό μέσο. Γενικώ είμαστε κανονισμένοι που το μέσο αυτό παρουσιάζεται με περισσότερη ευελιξία. Θα είναι προσανατολισμένο στην πολιτική μας και θα δώσει και την δυνατότητα οι πόροι να μπορούν να μεταφερθούν από ένα πεδίο πολιτικής σε κάποιο άλλο. Και οι χώρες θα έχουν πρόσβαση σε όλους τους τομείς πολιτικής ανεξάρτητα στο, από το σε, σε ποιο στάδιο της προταξιακής διαδικασίας βρίσκονται. Παρ' όλα αυτά, θέλω να ρωτήσω ορισμένα πράγματα. Θέλω περισσότερες λεπτομέρειες για το θέμα. Τώρα αρχίζουμε τις συζητήσεις, ετοιμάζουμε ε, ακροάσεις, αλλά ίσως από την αρχή θα έπρεπε να έχουν ξεκαθαριστεί μερικά πράγματα. Γνωρίζουμε Υπάρχει στην πρόταση δηλαδή της Επιτροπής το ότι πρέπει να ληφθούν ιδιαίτερα υπόψη πολιτικά κριτήρια, κυρίως στην περίπτωση των Δυτικών Βαλκανίων και οι ανάγκες των χωρών για το τι κάνουν με την ενίσχυση των θεσμών, με το δίκαιο, με την καταπολέμηση της διαφθοράς του οργανωμένου εγκλήματος, ε, τι γίνεται με την τήρηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων κλπ. κλπ είναι πράγματα και ειδικά, αλλά υπάρχουν και γενικά για την εκπαίδευση και πολλά άλλα. Τα θέματα αυτά αποτελούν κεντρικό πυλώνα της όλης διαδικασίας ένταξης. Οπότε, από αυτή την άποψη, οι τομείς πολιτικής που εντοπίζονται πώς αντικατοπτρίζουν τα κριτήρια αυτά ένταξης και κυρίως τις ανάγκες των χωρών αυτών στα Δυτικά Βαλκάνια. Και υπάρχει και ένα θέμα που πιστεύω ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διευκρινιστεί. Είναι το θέμα των τομέων πολιτικής, όπως αναφέρονται στον κανονισμό. Λέει ότι θα υπάρχει ένα μείγμα τομέων πολιτικής που θα αποφασίζεται από την Κομισιόν και τις ενδιαφερόμενες χώρες. Τι εννοείται όμως με αυτό σε ορισμένες περιπτώσεις κάποιοι μόνο τομείς πολιτικής ε, θα προσφέρονται ή σημαίνει το μείγμα αυτό ότι σε κάποιους τομείς πολιτικής θα υπάρχει πλήρης διάθεση, ενώ σε κάποιους άλλους λιγότερη, ότι θα επικεντρώνεται λιγότερο σε μερικούς τομείς πολιτικής ή ε, κομισιόν και σε άλλους περισσότερο. Τι ακριβώς σημαίνει αυτό. Ένα άλλο σημαντικό για μένα θέμα είναι το εξή. Δίνετε κάποιες απαντήσεις αρκετά γενικές για όλα τα μέσα, αλλά ειδικά για το προταξιακό μέσο, πώς βλέπετε το ρόλο τον ελεκτικό του Κοινοβουλίου. και όσον αφορά την πολιτική στρατηγική και τις επιμέρους στρατηγικές των χωρών. Θα ήθελα να ξέρω ποια είναι η άποψή σας προς το παρόν. Βέβαια, συνεχίζουμε να δουλεύουμε πάνω σε αυτό το θέμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Συνάδελφος Κούκαν στη συνέχεια και κατόπιν Μπραντνερ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Έχω δύο γενικές παρατηρήσεις και μετά θέλω να κάνω ορισμένες ερωτήσεις στους φιλοξενούμενους μας για να επωφεληθούμε από την παρουσία τους. Θεωρούμε ότι υπάρχουν κατευθυντήριες γραμμές σε αυτή τη δυνατότητα και ότι είναι βασικά τα ανθρώπινα δικαιώματα για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για τη συνεργασία με τις γειτονικές μας χώρες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται ένα μέσο το οποίο θα είναι αποτελεσματικό και θα τα αποκρίνεται στην πολιτική ηγητνιάσεως κατά τρόπον ώστε να στηρίξει ε, τις χώρες αυτές στις μεταρρυθμιστικές τους φιλοδοξίες. Θα πρέπει επίσης συγχρόνως να προχωρήσουν οι οικονομικές και πολιτικές μεταρρυθμίσεις και έχω να κάνω πέντε ερωτήσεις. Καταρχήν, σχετικά με την εφαρμογή της αρχής more for more. Δίνουμε περισσότερα για να πάρουμε περισσότερα. Πώς θεωρείτε ότι πρέπει να εφαρμοστεί στην πρακτική αυτή η ιδέα. Μπορείτε να μας πείτε ποιοι είναι οι οι δείκτες και οι μηχανισμοί παρακολούθησης σε αυτόν τον ε, κανονισμό και ποιες άλλες μορφές στηρίξεως μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε σε αυτή την προσέγγιση more for more. Επίσης, μπορούν να μας πούν σχετικά με την πρόοδο ποια ε, είναι τα, ε, οι τρόποι βαθμολόγησης της πρόοδου των χωρών αυτών σχετικά με τα κεφάλαια τα οποία δεσμεύονται για αυτές τις χώρες, πώς θα κατανεμηθούν μέσα στις χώρες αυτές εάν υπάρχει πλήρης σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τι, ποιος θα είναι ο ρόλος των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών στα πλαίσια αυτά. Ε, τη ε, θεωρούμε ότι θα πρέπει να ισχύσει η αρχή της αιρεσιμότητας και θετικά και αρνητικά. Ε, ποιοι είναι οι μηχανισμοί για να υπάρξει μία θετική αιρεσιμότητα και πώς πιστεύετε ότι μπορούμε να προωθήσουμε αυτή και την αρνητική αιρεσιμότητα διότι μέχρι στιγμής έχουμε δει πολλές περιπτώσεις όπου αυτό δεν έχει χρησιμοποιηθεί στην πολιτική γυκνιάσεως. Τέλος, ε, ε, πόσο πιστεύετε ότι πρέπει το, να διαμορφώσουμε τις πολιτικές μας προτεραιότητες. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Μπράννερ για τρία λεπτά. Yes, sorry, the microphone didn't work over there. Um, yes. Ναι, ευχαριστώ πρόεδρε. Θέλω να αναφερθώ στη δομή, στο πεδίο εφαρμογή και το δικαίωμα του Κοινοβουλίου για το μέσο σταθερότητα. Ε, μου αρέσει ότι το προηγούμενο άρθρο 4.3 ε, έχει ε, και η προετοιμασία έναντι των κρίσεων, έχει αναβαθμιστεί και επίσης μου, άρεσε το ότι η Κομισιόν πρότεινε να δαπανίσει το 65% του συνολικού προπολογισμού για την βραχυπρόθεσμη απάντηση της κρίσης. Εγώ θα ήθελα να αυξηθεί και στο 70% γιατί θεωρώ ότι η ικανότητα να απαντούμε σε κρίσεις είναι το πιο σημαντικό στοιχείο του μέσου για τη σταθερότητα και νομίζω θα μπορούσα να προσθέσω και κάποια ποσοστά για τα άρθρα 4 και 5 και θα πρότεινα 15 και 10% αντίστοιχα Δεύτερον, για το πεδίο εφαρμογή, θεωρώ ότι υπάρχουν πολλέ σημαντικέ τομεί πολιτική που δεν αναφέρονται στα τρία άρθρα και κυρίω στα παραρτήματα. Αλλά νομίζω ότι υπάρχουν κάποια πράγματα που θέλω να τονίσω και να αλλάξω θα ήθελα να ενδυναμώσω το συνδέσμο μεταξύ του οργανωμένου κλίματος και των πολιτικών καταπολέμησης της τρομοκρατίας, ε, κυρίως ό,τι αφορά την εφαρμογή, ε, μάλλον την παρακολούθηση του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο μέτρο Έχουμε επίσης ε, και την αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών. Χρειαζόμαστε πιο σαφή ορισμό σε αυτές τις περιπτώσεις. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το μέσο μόνο αν οι καταστροφές έχουν αντίκτυπο στη κατάσταση της ασφάλειας ε, και θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί το μέσο για να αντιμετωπίσουμε τις ανησυχίες της ασφάλειας που προκύπτουν από τις ε, ε, καταστροφές. Γιατί διαφορετικά έχουμε το ΕΚΟ και άλλα μέσα και για τον κοινοβουλευτικό έλεγχο. Τελευταίο σημείο υπάρχει ένα μεγάλο ερωτηματικό όπως και σε πολλά άλλα μέσα Δηλαδή, πιο ακριβώς θα είναι το δικαίωμά μας ως προς την άσκηση του ελέγχου ε, και εδώ συμφωνώ με άλλους ε, που ζήτησαν ε, ε της πράξης όπως και για άλλα μέσα και θέλουμε να ενδυναμωθεί το δικαίωμα του ελέγχου του Κοινοβουλίου για τα βραχυπρόθεσμα μέτρα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Μάριο Μάουρο, για το μηχανισμό εταιρικής σχέσης. Τρία λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Τρει σύντομε ερωτήσεις θέλω να απευθύνω συγκεκριμένα στους προσκεκλημένους μας. Βέβαια θα ήθελα να απαντήσουν και οι υπόλοιποι. Ε, θέλω να απευθυνθώ στον κύριο Μάρκ την περασμένη εβδομάδα στα πλαίσια μιας ανταλλαγής απόψεων με την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Ε, η κυρία Άστον ε, μας είπε ότι ο μηχανισμός εταιρικής σχέσης είναι ένας σαφής μηχανισμός εξωτερικής πολιτικής και θα έχει ένα κεντρικό ρόλο στην προώθηση των στρατηγικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά την άποψή σας, ποια είναι τα στοιχεία του μηχανισμού εταιρικής σχέσης που μπορούν να ενισχυθούν περαιτέρω για να υπογραμμίσουμε ακόμη περισσότερο τον κεντρικό ρόλο αυτού του μηχανισμού για την εξωτερική δράση της Ένωσης. Δεύτερη ερώτηση για τον ε, Διευθυντή, τον κύριο Ρούντι Σάουζερ το, ο μηχανισμός εσωτερική σχέσης απευθύνεται σε όλες αυτές τις χώρες ε, που ε, σχετίζονται με την εξωτερική δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, δηλαδή το μέσο έχει μια παγκόσμια επέκταση, με ποιους όρους μπορούμε να θεωρήσουμε ότι ο μηχανισμός εσωτερική σχέσης μπορεί να έχει ένα πρωταρχικό ρόλο σε σχέση με το μηχανισμό αναπτυξιακής συνεργασίας ό,τι αφορά τις χώρες της Λατινικής Αμερικής. Και η τρίτη ερώτηση για την ε, κυρία Μαρινάκη σε ποιο βαθμό και με ποιους όρους ε, ο μηχανισμός εταιρικής σχέσης πρέπει να απαντήσει σε απαιτήσει ταχείας επέμβαση σε σχέση με τις ε, τρίτες χώρες. Δηλαδή, ποιες είναι οι καταστάσεις που θα μπορούσαμε να φανταστούμε και ποια είναι η χρονική διάσταση για να μπορέσουμε να έχουμε αποτελεσματικές επεμβάσεις. Ευχαριστώ κύριε Μάουρο, σε ό,τι αφορά το μέτρο για τη δημοκρατία και τα ανθρωπίνα δικαιώματα, ο εισηγητής ε, λείπει, έτσι λοιπόν θα τον αντικαταστήσω εγώ, στο να θέσω τις ερωτήσεις που είναι τρεις. Καταρχήν, ε, δεν υπάρχουν κατεξουσιοδότηση πράξης ε, στην πρόταση αυτή. Αυτό αντίκειται στην ε, προσέγγιση που ακολουθήθηκε στην τελευταία συνδιαλλαγή. Έτσι λοιπόν έχετε δίκιο εσείς ε, για αυτό το γεγονός. Δεύτερον, ένα από τα σημεία κλειδιά αυτού του μηχανισμού θα έπρεπε να είναι η ευελιξία ε, πώς σκοπεύει η Κομισιόν και Υπηρεσία Εξωτερική Δράση να θέσει εφαρμογή την έννοια αυτή. Παραδείγματο χάρη στο μηχανισμό σταθερότητας, τρίτο σημείο και τελευταίο το μέσο για τα ανθρώπινα δικαιώματα και για τον εκδημοκρατισμό είναι να επικεντρώνεται κυρίως στα ανθρώπινα δικαιώματα και δεν εξετάστηκε η δυνατότητα να καταστεί ευρύτερη εντολή για τον εκδημοκρατισμό. Αυτές είναι οι ερωτήσεις ε, που έθεσα εγώ εκ μέρους ε, του κυρίου Λαμσπόρτοφ και Τώρα θα δώσω το λόγο σε κάποιον από τους, στον καθένα από τους ομιλητές. Έχετε στη διάθεσή σας 5-6 λεπτά για τις απαντήσεις και θα ξεκινήσουμε από την κυρία Μαρινάκη. Και κατόπιν θα ακολουθήσει ο Διευθυντής ο κύριος Σανίνο. Παρακαλώ. Thank you very much, Thank... Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε και ευχαριστώ πολύ για τη δυνατότητα που μας δίνατε συνάδελφοι και εγώ να βρισκόμαστε εδώ σήμερα μαζί σας. Ξεκινάει μια ανταλλαγή απόψεων, ένας διάλογος που θα μας οδηγήσει, ελπίζω, να καταλήξουμε στην, ε, στο πολιετές δημοσιονομικό ε, πλαίσιο και τα μέσα που περιλαμβάνει προκειμένου να στηριχθούν οικονομικά τα σχέδιά μας για το μέλλον. Κατά την άποψή μας πιστεύουμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να λάβουμε υπόψη μας τις παρατηρήσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου γιατί δίνουμε πολύ μεγάλη σημασία σε αυτά και στα σχόλια που θα ακούσουμε σήμερα στη συζήτηση. Πιο συγκεκριμένα τώρα για τα ειδικά μέσα, οι συνάδελφοι εδώ θα σας δώσουν όλες τις πληροφορίες που έχουμε. Τα διάφορα φόρουμς πάντως αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και να είσαστε σίγουροι ότι θα μελετήσουμε όλες τις δυνατότητες και όλες τις εναλλακτικέ λύσεις. Και σε αυτό είμαστε σίγουροι ότι εσείς μπορείτε να μας βοηθήσετε στο πολιτικό επίπεδο. Το πακέτο πάντως το οποίο καταλήξαμε πιστεύουμε ότι αντικατοπτρίζει τις προτεραιότητές μας για την ε, νέα δημοσιονομική περίοδο. Έτσι όπως ε, παρουσιάστηκαν στην ανακοίνωση για την Παγκόσμια Ευρώπη. Πιστεύουμε ότι αντικατοπτρίζουν επίσης τις σημερινές πολιτικές πραγματικότητες. Μεταξύ των διαφόρων μέσων, ποια είναι τα νέα στοιχεία τα οποία δεν υπήρχαν στις προηγούμενες περιπτώσεις τα προηγούμενα 7 χρόνια. Είναι αυτό μέσω εταιρικής σχέσης. Αυτό πραγματικά αποτελεί ένα νέο στοιχείο που έχουμε στη διάθεσή μας. Η πατή εκπρόσωπος και αντιπρόεδρος της Επιτροπής ήταν στην Επιτροπή σας, η κυρία Άστον, πριν από λίγο και είπε ότι πρόκειται για μια πρόσθετη αξία, γιατί για πρώτη φορά εξυπηρετούνται οι αξίες και οι στρατηγικές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. όπως για παράδειγμα η απάλληψη της φτώχειας. Το μέσο εταιρική σχέσης, λοιπόν, στο οποίο θα καταλήξουμε με τη δικιά σας την βοήθεια, γιατί οι ευρωβουλευτές θα βοηθήσουν να καταλήξουμε στην τελική μορφή, περιλαμβάνει διάφορα στοιχεία. Νέες, νέοι τομείς, νέες περιοχές συνεργασίας. Θα καλυφθεί ένα κενό Παρά το γεγονός ότι ο συνολικός, το ε, συνολικό ποσό δεν είναι τόσο μεγάλο, παρόλα αυτά θα αποτελέσει μία βάση για πολιτικές πρωτοβουλίες έτσι ώστε να προθίσουμε τον στρατηγικό μας σχεδιασμό και τις πολιτικές μας με εταίρους κλειδί απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κάτι το οποίο δεν κάναμε νωρίτερα γιατί έλειπε αυτό το μέσο. Συνεπώς, πρόκειται για ένα συμπληρωματικό ρόλο που θα συνδυαστεί με τα υπόλοιπα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας και έχουμε όλοι να αποφεληθούμε από αυτό. Όσον αφορά τώρα τον μηχανισμό για την πρόθεση της δημοκρατίας και τα ανθρώπινα δικαιώματα έχει αποδεχτεί, έχει αποδεχτεί ότι ήταν κάτι θετικό μέχρι τώρα. Δεν θα πρέπει εδώ να παραβλέψουμε κάτι το οποίο έχει λειτουργήσει τόσο καλά. Όλοι βέβαια βλέπουμε ότι κάτι θα μπορούσε να αλλάξει εδώ, κάτι εκεί, αλλά πρέπει να είμαστε προσεκτικοί να μην καταστρέψουμε ένα μηχανισμό ο οποίος έχει ως στόχο να προωθήσει τις αξίες μας προκειμένου να ενσωματωθούν σε όλες τις πολιτικές μας. Χαιρόμαστε που η διακυβέρνηση τώρα παίρνει τη θέση που της πρέπει σε έναν τομέα όπου πολλές χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν πολλά να κερδίσουν, έχουν πολλά να μάθουν. Είναι ένας τομέας ο οποίος έχει να κάνει και με την πρόθεση του παρατέρου διαλόγου για τα ανθρώπινα δικαιώματα, για την χρηστή διακυβέρνηση και όπου πιστεύουμε ότι κάθε κυβέρνηση μπορεί να προωθήσει και τις δικές της αξιολογήσεις για τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και αυτό θα ήταν ε, κάτι θετικό που θα ζητήσουμε. Η πολιτική μας θέλουμε να συμπεριλάβει όλους τους τομείς όπου πιστεύουμε ότι πρέπει να αναγνωριστεί η προσπάθεια που έχουν κάνει οι χώρες, ανεξάρτητα με το αν ήταν επιτυχής ή όχι οι προσπάθειες αυτές, αλλά αυτό πρέπει να αναγνωρίζεται έτσι ώστε να βοηθήσουμε με το δικό μας ε, μερίδιο στην προσπάθεια και με πιο στενή συνεργασία. Δεν θα ήθελα να σπαταλίσω περισσότερο το χρόνο σας. Οι συνάδελφοι τώρα να μιλήσουν και είμαι στη διάθεσή σας. Ευχαριστώ. Στέφανο Στέφανος Ανίνο έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον συνάδελφο για τα σχολεία του, κυρίω ε, επειδή υπογράμμισε ορισμένε από τι καινοτόμε ε, πτυχέ ε, για το προενταξιακό μέσο, για το μέσο προενταξιακή βοήθεια. Τώρα, να περάσω στι συγκεκριμένε ερωτήσει που τέθηκαν σε εμά σε ό,τι αφορά το θέμα τη εστίαση επί των πολιτικών κριτηρίων και ιδίω στου τομεί που σχετίζονται με το κράτο δικαίου. Αυτό είναι ακριβώς, μία, αυτή είναι μία από τις κεντρικές πτυχές ε, του μέσου προντοξιακής βοήθειας στον Οικονομισμό. Όπως γνωρίζετε, έχουμε προσδιορίσει, έχουμε εντοπίσει τα κεφάλαια 23 και 24 σε ό,τι αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα και την δικαιοσύνη ε, και ασφάλεια και είναι τα δύο κεφάλαια όπου θα πρέπει να αρχίσουμε τις επαφές και να εργαστούμε με τους πιθανούς υποψηφίους ακόμη και πριν την έναρξη των διαπραγματεύσεων. Ο Πρόκειται για τον πρώτο στόχο, για τον πρώτο χώρο πολιτικής και το πλαίσιο όπου θέλουμε να υποστηρίξουμε περισσότερο το θεσμικό πλαίσιο των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων. Μία από τις αδυναμίες που εντοπίσαμε στο ΙΠΑ 1, στο πρώτο κανονισμό, είναι ακριβώς ότι η υποστήριξη που δίναμε στην οικοδόμηση θεσμών, ε, των θεσμών που σχετίζονταν με την ε, διαχείριση της βοήθειας των ε, ταμείων για τη γεωργία και την απασχόληση, ίσως να μην κάλυπτε επαρκώς το θέμα του κράτου δικαίου και θέλουμε τώρα να διασφαλίσουμε ότι αυτό διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στην δραστηριότητα που πρόκειται να αναπτύξουμε και να διασφαλίσουμε ότι η βοήθεια μπορεί να υποστηρίξει τη διαδικασία αυτή. Δεύτερη ερώτηση αφορά τους τομείς της πολιτικής και το μείγμα. Προσπαθήσαμε να ξεπεράσουμε τη διάκριση μεταξύ των διάφορων συνιστοσών των, του μέσου όσο έχει αυτή τη στιγμή και να προσδώσουμε μεγαλύτερη ευελιξία. Θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι δεν θα έχουμε μία προσέγγιση, ένα μέγεθος τερνιάζει σε όλα, αλλά διαφορετική προσέγγιση ε, που θα εξετάζει τις συγκεκριμένες ανάγκες και ικανότητες της κάθε χώρας και που θα μπορεί να εξετάσει και τα διάφορα στάδια στη διαπραγματευτική διαδικασία έτσι ώστε να μπορέσουμε να προσδώσουμε το κατάλληλο μείγμα της βοήθειας ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε χώρας προσπαθούμε, και αυτό είναι το άλλο σημαντικό στοιχείο, να απομακρυνθούμε από ε, κάποιου είδους απομονωμένα κονδύλια που θα έχουν εκταμιευτεί εκ των προτέρων και θέλουμε να βρούμε τρόπους να συμφωνήσουμε επί μια στρατηγική εναντί των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων ε, και να καθορίσουμε το μείγμα πολιτικής βάση των συγκεκριμένων αναγκών. Και πάλι νομίζω ότι είναι προφανές ότι αυτό που χρειάζεται, το χάρη, για μια χώρα που ξεκινά τις διαπραγματεύσεις ε, για την προσχώρηση, ε, δεν είναι ίδιες οι ανάγκες αυτής της χώρας με τις ανάγκες μια χώρας με την οποία ξεκινάμε τώρα τη μελέτη σκοπιμότητας για συμφωνία σταθερότητας και σύνδεση, όπως το κοσφοπέδιο, το χάρη. Και η τρίτη σα ερώτηση, ό,τι αφορά τον έλεγχο, το ρόλο ελέγχου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και την εμπλοκή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, νομίζω ότι αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να ειδωθεί υπό το ευρύτερο πρίσμα των συζητήσεων με την ε, Κομισιόν καλύπτεται και άλλα οριζόντια θέματα που έχουν να κάνουν με τα, εξωτερικά, με τα μέσα εξωτερική δράση, ό,τι αφορά το ΙΠΑ, το μέσο προενταξιακή βοήθεια. Αυτό που μπορώ να πω βάσει του νέου κανονισμού επιτροπολογία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα λάβει όλα τα σχέδια των εγγράφων ε, τη στιγμή που θα στέλνονται και στα μέλη της Επιτροπής ΙΠΑ και στο στάδιο αυτό, αυτό που μπορώ να προσθέσω και Επίση, ε, θα ήθελα να δω την εντατικοποίηση των σχέσεων ε, μεταξύ του Επιτρόπου Φίλου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των ε, βουλευτών. Είναι το ότι πέρα από το νομικό πλαίσιο, σίγουρα είμαστε ανοιχτοί στο να κάνουμε μια τακτική και σβάθος ανταλλαγή απόψεων προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα εγκρίνει ε, τις αποφάσεις και τους προσανατολισμούς που λαμβάνουμε. Αλλά και πάλι υποθέτω ότι αυτό θα είναι ένα στοιχείο που θα πρέπει να ειδωθεί σε ένα ευρύτερο πλαίσιο. Έτσι λοιπόν δεν θα ήθελα να αναφερθώ περαιτέρω στο στάδιο αυτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ εγώ εσάς και επειδή σεβαστήκατε και το χρόνο. Τώρα το λόγο έχει ο κύριος ε, Ρούντι Σάουρ, παρακαλώ. Thank you, Chairman. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για την, για την ευκαιρία που μου δίνετε για αυτή την ανταλλαγή και πρέπει να χαρακτηρίσω το πακέτο με τέσσερις φράσεις γιατί ε, έτσι θα απαντήσω σε πολλές ερωτήσεις που έχουν τεθεί. Πρέπει δηλαδή να καταλάβουμε ποια είναι ε, η λανθάνουσα συλλογιστική αυτού του πακέτου. Έχει καταρτιστεί από όλε τις Επιτροπές Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ε, έχει παρουσιαστεί ή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι τα μέσα έχουν συντονιστεί και υπάρχει καλύτερη δυνατή, ο καλύτερος δυνατός καταμερισμός του χρόνου μεταξύ των διαφόρων μεθόδων. Θα επανέλθω στο σημείο αυτό. Και επιπλέον υπάρχει ένα νέο στοιχείο απλοποίησεως για την εφαρμοστική νομοθεσία η οποία θέτει τους ίδιους κανόνες για όλους και αυτό είναι σημαντικό για διάφορα θέματα που έθεσαν ε, τα μέλη αυτής της Επιτροπής. Το επόμενο είναι ότι το πακέτο αυτό αντικατοπτρίζει ακριβώς την συνθήκη της Λισαβόνας και σε κάθε περίπτωση αναφερόμαστε σε ένα τομέα που αναφέρεται εις την συμφωνία και οι αλλαγές είναι εσωτερικές μέσα στα διάφορα μέσα και εκεί ε, έχουμε από επιζητήσει την απλοποίηση του κάθε ε, μέσου και αυτό έχει λεχθεί. Ένα βασικό θέμα λοιπόν είναι ότι ε, το πακέτο αυτό και το ποσό στο οποίο βασίζεται είναι ο μόνος τομέας όπου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε αύξηση της χρηματοδοτήσεως, δηλαδή πριμοδότησε την χρηματοδότηση της εξωτερικής δράσης μέσω αυτού του πακέτου. Ε, ορισμένα θέματα δεν αναφέρθηκαν και εδώ θα αναφερθώ τώρα στην ερώτηση του κυρίου Κουκάν. Πρέπει να εξετάσουμε το θέμα σαν ένα σύνολο και βλέπουμε ότι εδώ υπάρχει ε, εμπλοκή της ε, κοινωνίας των πολιτών των πολιτών, κατανομή των ε, πόρων, ε, διάφοροι τρόποι με τους οποίους προσπαθούμε να επιτύχουμε καλύτερη συνεκτικότητα στην εξωτερική μας δράση, διότι πολλές φορές εφαρμόσουμε διάφορα μέσα συγχρόνως, αλλά με κάποιο βάσιμο λόγο. Ε, και γι' αυτό Όλα αυτά έχουν ε, θεωρηθεί σε κάθε περίπτωση σαν μία δυνατότητα και δεν διατίθενται εκ των προτέρων όλοι οι πόροι κατά τρόπον ώστε να διατηρηθούν ορισμένα αποθέματα σε περίπτωση ανάγκης. Πράγμα το οποίο μέχρι στιγμής χρειαστήκαμε μόνο στο Ευρωπαϊκό ε, Ταμείο Ανάπτυξης όσον αφορά την ερώτηση του κυρίου Μάουρο. Πρέπει να είμαστε σαφείς. Ο στόχος ε, του μέσου ε, συνεργασίας δεν είναι να καταστεί ένα μέσο ανάπτυξης, ιδίως για τις χώρες της Λατινικής Αμερικής. Για ορισμένες χώρες της Λατινικής Αμερικής προτείνουμε μία νέα συνεργασία αλλά η DCI θα είναι ο βασικός αγωγός μας και δεν θα λογιστεί αυτή η ενίσχυση σαν αναπτυξιακή για να μπορέσουμε να αυξήσουμε τις δυνατότητες συνεργασίας. Ε, όσον αφορά την Βάιστα, ε, νομίζω ότι πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι κινούμαστε σε ένα γενικό πλαίσιο και υπάρχουν ε, ορισμένες πράξεις ε, όπου κατά την εφαρμογή θα αλλάξουν οι προτεραιότητες ή η προσέγγιση και θα χρειαστούμε κατεξουσιοδότηση πράξεις οι οποίες ε, θα ενισχύσουν το μέσο ανάπτυξης Γι' αυτό και δεν προβλέπουμε να αλλάξουμε σημαντικά την, ε, ορισμένα μέτρα κατά την ανάπτυξή τους, αλλά αλλού έχουμε αυτές τις δυνατότητες. Και τέλος ε, το ερώτημα του κυρίου Λάμστορφ. Πρέπει να σας πω ότι ο εκδημοκρατισμός λαμβάνεται υπόψη σε όλα τα μέσα και όχι μόνο στο μέσο για τον εκδημοκρατισμό ε, γιατί θα ήταν κρίμα. Είτε μιλάμε για ανάπτυξη, είτε για εκδημοκρατισμό, είτε για επενδύσεις ε, ε, τονίζουμε περισσότερο τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις διαδικασίες τις εκλογικές για να υπάρξει ταχύτερη πρόθεση της, του εκδημοκρατισμού. Ο κύριος Μάρκ έχει το λόγο. Να απαντήσω πρώτα στις ε, ερωτήσεις της κυρίας Μπράντρες σχετικά με τον ε, μηχανισμό του δημοσιονομικού πλαισίου. Την ευχαριστώ πολύ πάντως για τα διάφορα στοιχεία που μας έδωσε όσον αφορά την βελτίωση του ΕΦΕΣ. Είναι αλήθεια ότι αυτό που προσπαθούμε να πετύχουμε είναι να διασφαλίσουμε ότι υπάρχει περισσότερη ελαστικότητα αλλά και ταχύτητα προκειμένου να έχουμε αποτελέσματα βραχυπρόθεσμα. Είναι αλήθεια όμως επίσης ότι έχουμε επιμείνει ότι θέλουμε βελτίωση και στις μακροπρόθεσμες δυνατότητες για να αποφεύγονται κρίσεις, για να υπάρξει οικοδόμηση ειρήνης κλπ. Τώρα θέλω να προσθέσω ότι όσον αφορά τις προτάσεις της για το ότι πρέπει να βγάλουμε από το εύρος εφαρμογής του μηχανισμού τα στοιχεία που έχουν να κάνουν με φυσικές καταστροφές, εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει να διατηρηθεί το εύρος εφαρμογής. Και αυτό είναι γιατί η ΕΚΟ μπορεί να παρέμβει αμερόληπτα για να ε, βοηθήσει σε περίπτωση φυσικής καταστροφής, αλλά αυτό που δεν μπορεί να κάνει είναι να φτάσει στην ρίζα του κακού, που μερικές φορές έχει πολιτικές διαστάσεις. Επίσης, πιστεύουμε ότι το ΕΦΕΣ μπορεί να καλύψει το κενό ανάμεσα στην ανακούφιση και την ανοικοδόμηση. Είναι κάτι που χρειάζεται σε οποιαδήποτε περίπτωση παρέμβασης μετά από κάποια φυσική καταστροφή. Είναι πολύ βασικό αυτά τα στοιχεία να τα έχουμε αν θέλουμε να αναπτύξουμε σχεδιασμό και να έχουμε μια μακροπρόθεσμη απάντηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα θέλουμε τα εύρος εφαρμογής να μείνει ως έχει. Τώρα για το θέμα που έθεσε ο κύριος Μάουρο, για το τι στοιχεία θα μπορούσαν να ενισχυθούν παρετέρω σε σχέση με το PI, ώστε να προσανατολίσετε περισσότερο στην πολιτική. Πιστεύουμε ότι η τρέχουσα πρόταση παρουσιάζει μια καλή ισορροπία ανάμεσα στους στόχους που είναι η διεθνής διάσταση της Ευρώπης 2000 και να αντιμετωπιστούν και μεγάλες προκλήσεις. Κυρίως χρειάζεται διάλογος για θέματα όπως είναι οι κλιματικές αλλαγές και η ενέργεια. Ο δεύτερος στόχος που έχει να κάνει με την βελτίωση της πρόσβασης στην αγορά και περισσότερες ευκαιρίες εμπορικές για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις είναι κάτι που πρέπει να διατηρηθεί. Αλλά δεν είναι ζωτική σημασία. Ο κύριος στόχος είναι αυτός που ανέφερα νωρίτερα. Είναι ένας μηχανισμός προσανατολισμένος στην εξωτερική πολιτική. Το θέμα τώρα της προβολής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην παγκόσμια σκηνή μέσω της διπλωματίας, της ακαδημαϊκής συνεργασίας, της εκπαίδευση κτλ. έρχεται σε τρίτη θέση. Με δύο λόγια δηλαδή, πιστεύουμε ότι η πρόταση είναι καλά ισορροπημένη και ότι αντικατοπτρίζει τους κύριους στόχους του PI, που είναι ακριβώς ένας χρήσιμος μηχανισμός που δεν είχαμε μέχρι τώρα και που πρέπει να αναπτύξουμε παρετέρω. Ευχαριστώ. Thank you. Ευχαριστώ. Η κυρία Γκόμες, δύο λεπτά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και όλους τους εκπροσώπους από τις ε, υπηρεσίες της Κομισιόν που μας έδωσαν πληροφορίες και την υπηρεσία εξωτερικής δράσης. Ε, δεν καταλαβαίνω γιατί δεν έχουμε μία κοινή γλώσσα σε όλα τα μέσα, σε όλους τους μηχανισμούς, γιατί δεν έχουμε μία κοινή εφαρμοστική διαδικασία και κοινού εφαρμοστικούς κανόνες. Νομίζω ότι θα έπρεπε να στοχεύσουμε σε η μεγαλύτερη εναρμόνιση των διαφορών μέσων. Φυσικά θα συνεχίσουν να υπάρχουν ιδιαιτερότητες και θα γίνεται ξεχωριστή διαπραγμάτευση, αλλά θεωρώ ότι πρέπει να τα διατηρήσουμε ως πακέτο, όπως υπόθηκε, και προκειμένου να προσπαθήσουμε να εναρμονίσουμε εναρμονίσουμε ό,τι μπορεί να εναρμονιστεί και θα έπρεπε να εναρμονιστεί. Και θα έπρεπε να εναρμονιστεί ο θεσμικός ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Νομίζω ότι το Κοινοβούλιο πρέπει να έχει ένα ρόλο στον προγραμματισμό και στο στάδιο της εφαρμογής. Έτσι λοιπόν ε, το θέμα των κατεξουσιοδότηση πράξεων είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα και θα πρέπει να είναι ε, ουσιαστικά ένα νήμα που θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε και είναι πραγματικά πολύ σημαντικό ο ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ορισμένες διαδικασίες δίνονται ω αρμοδιότητε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δηλαδή όχι μόνο για την πρόθεση των δραστηριοτήτων, αλλά και για διαβουλεύσει. Θα πρέπει να προβλέπετε και αυτό. Και επίση ε, θεωρώ ότι θα πρέπει αυτό το σύνθημα περισσότερο και περισσότερο θα πρέπει να είναι κάτι περισσότερο από σύνθημα, αλλά πραγματικότητα. Θα πρέπει να γίνει πραγματικότητα σε όλους τους μηχανισμούς και φυσικά θα πρέπει να υπάρχει αιρεσιμότητα στην παροχή της βοήθειας και θα πρέπει να γίνεται διάκριση μεταξύ των κυβερνήσεων, παραδείγματος χάρη. Ε, που δεν συνεργάζονται και δεν ε, κινούνται προς τον εκδημοκρατισμό και το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ε, δηλαδή, όχι να σταματάμε τη χορήγηση των πόρων, αλλά να χορηγούμε τους πόρους, να τους διοχετεύουμε στις χώρες που ακριβώς αγωνίζονται υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θα έλεγα ότι ο τρόπος που έχει δοθεί η βοήθεια μέχρι τώρα είναι αρνητική και δεν ε, συνάδει με την προσέγγιση more for more, περισσότερα για περισσότερα. για το μέσο DCI, το Μηχανισμό Αναπτυξιακής Συνεργασίας. Ε, κάποια που είπα φυσικά ισχύουν και για το Μηχανισμό Αναπτυξιακής Συνεργασίας και θέλω να ρωτήσω τι γίνεται με το EDF, ε, γιατί μιλάμε για το DCI και λέμε ότι ε, αφορά όλες τις χώρες ε, σκοπεύει αυτός ο μηχανισμός στην εξάλληψη της ανέχειας και υπάρχουν και άλλοι στόχοι όπως η πρόθεση της δημοκρατίας, του κρατούς δικαίου κτλ αλλά ε, μιλάμε για ένα μεγάλο ποσό κονδυλίων που πηγαίνουν μέσω του DF και δεν υπάρχει προϋπολογισμός. Ε, γιατί δεν εκπονείται προϋπολογισμός για το μέσο αυτό και να υπάρχει δημοκρατικός έλεγχος. Γιατί δεν χρησιμοποιείται λοιπόν για να καλυφθούν οι χώρες ε, τις οποίες δεν έχουμε συγκεκριμένη σχέση. Και διακόπτεται το μικρόφωνο της ομιλήτριας. Δεν ακούμε πια τη λέει Τέλος, θέλω να θέσω μια ερώτηση. Ποια είναι η δυνατότητα να δούμε κατεξουσιοδότηση πράξης σε ό,τι αφορά το Ευρωπαϊκό Μέσο για τη Δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα, δηλαδή ε, να υπάρχει ερωγή και τη Επιτροπή για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τον Εκδημοκρατισμό. Τι είναι αυτή η Επιτροπή, γιατί είδα αυτή την Επιτροπή να αναφέρεται σε κάποιο από το έγγραφα. Ματ Λένερ, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα μπορούσα να μιλήσω και τα λεπτά παραπάνω από την προλαλή σας. Θα προσπαθήσω όμως να είμαι σύντομος. Όλα αυτά ακούγονται πάρα πολύ ωραία, πολύ καλά σχέδια αλλά βλέπουμε ένα κατάλογο επιθυμιών. Περισσότερα χρήματα να δίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Κοινοβούλιο. Αλλά διαπραγματευόμαστε λιγότερα χρήματα για την Ευρωπαϊκή Ένωση την ίδια. Οπότε τα χρήματα αυτά από πού έρχονται. Πού βρεθήκαν αυτά τα χρήματα. Για να κάνει κανείς σχέδια χωρίς όριο είναι εύκολο, αλλά δεν είναι καθόλου λογικό. Ρωτώ λοιπόν, Επιτροπή και Κοινοβούλιο, από πού έρχονται αυτά τα χρήματα, Πώς είσαστε σίγουροι ότι υπάρχουν αυτά τα χρήματα και ποιο, ποια άλλη δαπάνη θα χάσει για να βρεθούν αυτά τα χρήματα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ζητήσει να ξοδεύει λιγότερα χρήματα. Αυτό θέλουμε. Η Ολλανδία, η Αυστρία, η Δανία, η Γερμανία, η Γαλλία, ένα σωρό χώρες ζήτησαν εξοικονόμηση πόρων. Να ξοδεύουμε λιγότερα. Όλοι. Η Ολλανδία, για παράδειγμα, 2 δισεκατομμύρια λιγότερο θα δαπανίσει. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει και αυτή να προσαρμοστεί και να συνηθίσει στην ιδέα ότι πρέπει λιγότερα να ξοδεύει και όχι περισσότερα. Είναι πολύ περίεργο λοιπόν να βλέπουμε εδώ πέρα και να συζητάμε για τόσα εκατομμύρια που θα δαπανηθούν σε όλα αυτά τα προγράμματα, ενώ από την άλλη μεριά πρέπει να εξοικονομήσουμε πόρους. Μετανάσταση, για παράδειγμα, έρχονται από τόσο φτωχές χώρες στην Ευρώπη και δημιουργούν ένα σωρό προβλήματα μεταξύ άλλων που ισλαμοποιούνται οι χώρες μας. Όλα αυτά πρέπει να τα σταματήσουμε. οι χώρες αυτές που σας είπα πριν ζητάνε περισσότερα χρήματα στη Frontex για να ελέγχουμε τους ελέγχους μας. Λοιπόν, απαντήστε μου, πού βρίσκονται αυτά τα χρήματα. Η προηγούμενη μίλησε τρία λεφτά παραπάνω. Γιατί εγώ όχι, Πρόεδρε. Δεν κόψατε την προηγούμενη ομιλήτρια και κόβετε εμένα. Γιατί. Ευχαριστώ. Λέει Εσείς έχετε δίκιο όταν ζητάτε σεβασμό του χρόνου. Γιατί, κοιτάξτε, θέλουμε να σεβαστούμε και τους συνάδελφους που θα ακολουθήσουν συνέχεια και έχουν τα ίδια δικαιώματα. Δώσαμε λίγο παραπάνω χρόνο στη συνάδελφο Γκόμες γιατί είναι συγγήτρια. Και αυτός ήταν ο λόγος για τον οποίο είχαμε κάποια ανοχή. Όμως είμαστε σίγουροι ότι η κυρία Γκόμες θα προσέχει ε, στη συνέχεια και θα σέβεται το χρόνο. Επόμενος ομιλητής. Ε, ε, Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Αδαμανάκη. Παρακολουθήσαμε την ε, ο ε, Μαρινάκη. Ε, παρακολουθήσαμε με ενδιαφέρον αυτά που είπατε και ε, πρέπει να προωθήσουμε τις ευρωπαϊκές αξίες και να αναβαθμίσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή η ανάλυση λοιπόν ήταν πολύ εκτενής που έγινε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θέλω να σας πω κάτι το οποίο όμως με ενόχλησε ότι ένα από τα καλά μέσα που είναι ε, το μέτρο της ε, βορείας ε, διάστασης όπου μιλήσαμε για τη Βόρειο Θάλασσα αλλά φοβάμαι ότι τώρα εάν μεταφερθεί αυτή η χρηματοδότηση για τη Βόρειο Θάλασσα ή στη συνεργασία θα μειωθεί στον άλλο τομέα η χρηματοδότηση πράγμα το οποίο σημαίνει ότι δεν θα έχουμε επαρκή χρηματοδότηση για την βόρεια διαστασία η οποία έχει λειτουργήσει πολύ καλά μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και της Ρωσίας και υπάρχει και ε, μία συνεργασία μεταφορών στην, με αρκτική διάσταση. Θέλω λοιπόν να ρωτήσω, θα επαρκέσει η χρηματοδότηση ή όχι υπό αυτά τα συνθήκε. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ που δώσατε και το χρόνο. Λοιπόν, συνάδελφος Κάτσεν, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα μιλήσω εκ μέρους της πολιτικής μου ομάδας και θέλω να πω κάτι για το ύπνο. Όταν ολοκληρώνει η χώρα μου την διαδικασία της προσχώρησης, ε, ποτέ δεν είχαν, υπήρχαν κάποιοι που δεν είχαν ακούσει το πρόγραμμα ε, και ε, στη συνέχεια όμως διαδόθηκε και έγινε τόσο γνωστό όπως το Εράσμους. Τώρα όμως όταν μιλάω σήμερα σε συνεργάτες μου στα Δυτικά Βαλκάνια, σε συνομιλητές μου, μου λένε ότι project που έχουν ε, χορηγό την Κίνα, παραδείγματος χάρη, έχουν μεγαλύτερη προβολή από αυτά που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και μάλιστα ακόμη και αν τα κινέζικα έργα δεν είναι τόσο σχετικά με την ανάπτυξη της υποδομής με την θεώρηση του ΙΠΑ πρέπει να αυξήσουμε την προβολή και τη ευρωπαϊκή χρηματοδότηση αλλά και τη διαδικασία προσχώρηση αυτή καθ' αυτή. Ε, στη βελτίωση της καθημερινή ζωή ε, των πολιτών, ε, των χωρών ε, προσχώρησης ε, το ΙΠΑ θα πρέπει να συνεισφέρει στην βελτίωση της ποιότητας ζωής και των συνδικών εργασίας και θα έπρεπε να γίνει αυτό με έναν τρόπο που το σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, να είναι σφραγίδα σε όλη τη διαδικασία. Επίσης πρέπει να συνδέσουμε την δημιουργία με την εφαρμογή των στόχων καθώς συχνά συμβαίνει οι βελτιώσεις να λαμβάνουν χώρα αλλά μόνο στα χαρτιά και όχι στην πραγματική ζωή σας. Ευχαριστώ. Πολύ ωραία. Παρακαλώ, κυρία Νίνσκι. Ευχαριστώ, αγαπητοί συνάδελφοι. Ως σκιώδης εισηγητρία για το ΕΛΚ, ε, για την πρόταση για το πρωτοξιακό μέσο, μέσω παραδοξιακής βοήθειας, ε, θέλω να ευχαριστήσω τους εκπροσώπους της Κομισιόν και της ε, ΙΕΔ για την συνεισφορά τους στη συζήτηση για την πρόταση του IPA πιστεύω ότι πρέπει να επικεντρωθούμε σε τρία κυρία ζητήματα. Καταρχήν χρειαζόμαστε μεγαλύτερη σαφήνεια στη σύνδεση των στόχων ε, του μέσου με του συγκεκριμένου δείκτες για τη μέτρηση τη πρόοδου. Δεύτερον, πρέπει να δημιουργήσουμε σαφή σύνδεσμο μεταξύ τη πρόοδου που έχουν πετύχει δικαιούχοι και τι ε, ε, τελικές ε, τα τελικά κονδύλια που λαμβάνουν. Επίση, πρέπει να υπάρχει συνέπεια όχι μόνο ε, μεταξύ του αλλά του EPA και του χρηματοδοτικού κανονισμού και τέλος ε, θα εκτιμούσα εκπρόσωποι της Κομισιόν και της ε, Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης να σχολιάσουν κάποια σημεία. Καταρχήν, μια πιθανή δημιουργία ενός αποθεματικού ε, επιδόσεων που μάλλον των έργων που έχουν χρησιμοποιηθεί τα κονδύλια, πώς θα διαφοροποιήσετε μεταξύ της καλής και της κακής εκτέλεσης και τρίτον θα σκεφτόσαστε να χρησιμοποιήσετε τα ε, κονδύλια earmarking ε, θέτοντας ε, ονομαστικούς όρους και τέλος θα χρησιμοποιούσατε άλλους δείκτες πέρα από τις κατανομένες ονομαστικούς όρους για να λάβετε υπόψη το μέγεθος της οικονομίας της δικαιούχου χώρας όταν λαμβάνετε υπόψη την αλλαγή της χρηματοδότησης του κάθε μηχανισμού σε τρέχουσες τιμές, πόσες χώρες έχουν αναπτυχθεί και θα έχουν αναπτυχθεί μέχρι το έτος 2020 και ο αριθμός των συμπεριλαμβανομένων χωρών, η αυξημένη χρηματοδότηση δεν είναι τόσο μεγάλη όπως την παρουσιάσετε κυρία Ρούντις Χάουσερ. Ευχαριστώ. Μπραντνερ, δύο λεπτά. I didn't need minutes. Δεν θέλω δύο λεπτά. Θέλω μόνο να απαντήσω σε σχόλιο που έγινε για τις φυσικές καταστροφές. Είναι ενδιαφέρουσα απάντηση που δώσατε. Είπατε ότι είναι και το θέμα της ρίζας, της πηγής. Ναι, αλλά φυσικές καταστροφές τι πηγή έχουν, τι ρίζα έχουν. Οι σεισμοί, πώς μπορούμε να καταπολεμήσουμε την πηγή. Ή όταν οι άνθρωποι προκαλούν ε, καταστροφές, αυτές ε, συνήθως παίρνουν πάρα πολύ χρόνο για να φτάσουμε εκεί. Και δεν ξέρουμε από πριν πότε θα γίνουνε. Να μιλάμε γενικά για φυσικές καταστροφές ή για καταστροφές που προκαλούν ε, οι άνθρωποι, μου φαίνεται ότι δεν θα πρέπει έτσι γενικά να βάζουμε λεφτά. Όταν υπάρχει για κάτι συγκεκριμένο, για να προλάβουμε ε, κάποια καταστροφή που οφείλεται σε έλλειψη ασφάλειας, τότε ναι. Κατά τα άλλα δεν πείθομαι. Ε, για δύο λεπτά παρακαλώ. Ε, Ευχαριστώ. Είμαι η συγγήτρια, συντάκτρια μάλλον γνωμοδότησης για το Μηχανισμό Σταθερότητας και Δημοκρατίας και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Εδώ είμαι η η συγγήτρια για το Μηχανισμό Εταιρικής Σχέσης. Πιστεύω λοιπόν ότι είναι πολύ σημαντικά αυτά που είπαν διάφοροι προλαλήσαντες εδώ για το ότι πρέπει να υπάρχει συνεργασία όλων των μηχανισμών για να μην τρελαθούμε από τους διαφορετικούς μηχανισμούς και διαφορετικές παραμέτρους για τον καθένα από το μηχα... τους μηχανισμούς αυτούς. Έχω κάποιες συγκεκριμένε ερωτήσεις. Πρώτον, σε σχέση με τον μηχανισμό για τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αναφέρθηκε, το είπατε εσείς και ο κύριος Λάμπστορφ, ότι επικεντρώνεται στα ανθρώπινα δικαιώματα κυρίως και λιγότερο στη δημοκρατία. Θα ήθελα να διευκρινιστεί ποια είναι η χρηματοδότηση του Democracy Endowment που εγκρίθηκε με κονδύλια αυτού του μηχανισμού και που θα ζητήσουμε από την Επιτροπή Προπολογισμών. Δεύτερον, ο μηχανισμός που έχει να κάνει με την εταιρική σχέση. Από αυτά που είπε η Επιτροπή κατάλαβα ότι πρόκειται μεταξύ άλλων και για κονδύλια για εξαγωγές, δηλαδή πώς θα βοηθήσουμε τρίτες χώρες να αγοράζουν ευρωπαϊκά προϊόντα. Μπορείτε παρακαλώ να μου το διευκρινίσετε αυτό, έτσι είναι ή όχι. Τρίτον, σε σχέση με το μηχανισμό σταθερότητας, με την κυρία Μπράντον δουλεύουμε πάνω σε αυτό και παρακολουθούμε την ε, ε, χρήση των πόρων. Συμφωνούμε τις περισσότερες φορές σε αυτήν, όμως στην περίπτωση η κυρία Μπράντερ λέει ότι θα ήθελε το 70% των κοδηλίων να πηγαίνουν σε μη προγραμματισμένες δράσεις, δηλαδή έκτακτες, και θα ήθελε εδώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μου πει στην πραγματικότητα τι χρειάζεται, 35% των κονδυλίων για την προγραμματισμένη βοήθεια. Είναι το ελάχιστο, αναγκαίο, για να χρησιμοποιηθεί το τμήμα εκείνο του μηχανισμού που πάει στην προγραμματισμένη βοήθεια και όχι στην έκτακτη. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ελαφράγκα για το κλείσιμο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Χαίρομαι πάρα πολύ που έχουμε αυτή την ενδιαφέρουσα συζήτηση για τα χρηματοδοτικά μέσα, ε, δυνάμει των δημοσιονομικών προοπτικών ε, και χαίρομαι που θα υπάρχει διαφοροποίηση καταρχήν ε, στο μέσο για την γειτονία και για την αναπτυξιακή βοήθεια. Έχω δύο ερωτήσεις για το μηχανισμό γειτονίας πώς ε, θα θεσπιστεί η αρχή more for more που ουσιαστικά είναι το κύριο στοιχείο που διέπει όλη αυτή τη συζήτηση γιατί σε ό,τι αφορά την παρακολούθηση των διαδικασιών μετάβασης ε, των χωρών της Αραβικής Άνοιξης όλο αυτό δεν λειτουργεί πολύ καλά και με ανησυχεί και Πρόεδρε το θέμα του μηχανισμού αναπτυξιακής βοήθειας και υπάρχει ε, η διαφοροποίηση αλλά εδώ έχουμε 17 χώρες μέσα... Εισοδήματο και δύο χώρες ε, χαμηλού εισοδήματο και πολλές από αυτές βρίσκονται και στη Λατινική Αμερική και σε όλο αυτό το εγχείρημα θα χάσουν πολλά χρήματα. Αυτή τη στιγμή το Κοινοβούλιο είναι έτοιμο να κυρώσει τη συμφωνία με το Περού και με την Κολομβία και το να από τις χώρες αυτές ε, ε, το, και από το Κουαδόρ αυτό το μέσο είναι κάτι αδέξιο γιατί στη Λατινική Αμερική συνεχίζουν να υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλε ανισότητε και νομίζω ότι πρέπει να δούμε πώ θα λύσουμε αυτό το πρόβλημα. Πρέπει να λάβουμε υπόψη την κοινωνική συνοχή, τι απειλέ κατά τη διαδικασία εκδημοκρατισμού, γιατί 140 εκατομμύρια άτομα σε αυτή την ε, υποήπειρο ε, ζουν σε ανέχεια. Έχουμε πολλά εκατομμύρια που δεν έχουν πρόσβαση στην υγεία και 10 από τι χώρε τη Λατινική Αμερική ε, βρίσκονται στην πιο, σε κατάσταση κατάσταση ε, Στο Σαντιάγο της Χιλής είπαμε ότι θα ε, ε θα προβοηθήσουμε αυτή την ε, Ήπειρο να οικοδομηθεί, όμως εδώ δίνουμε το λάθος μήνυμα. Ναι, να έχουμε αρχή διαφοροποίησης, αλλά να προσπαθήσουμε να δούμε και ποιες είναι οι περιστάσεις και πώς πρέπει να τις σεβαστούμε. Σε αυτό το σημείο να δώσουμε το λόγο στους ομιλητές και τους παρακαλούμε να απαντήσουν στις ερωτήσεις ε, που έχουν τεθεί από τους συναδέλφους και να σας υπενθυμίσω και τις ερωτήσεις που τέθηκαν και από μένα στην αρχή. Ιδίω σε ό,τι αφορά του τρόπου συνεργασία που θα εφαρμοστούν ε, μεταξύ τη Υπηρεσία Εξωτερική Δράση και τη Κομισιόν ε, στα διάφορα προγράμματα. Δεύτερον, ποιοι μηχανισμοί συντονισμού προβλέπονται με του άλλου δωρητέ. Και τρίτον, ποιοι τρόποι διαλόγου θα λάβουν χώρα με τι χώρε εταίρου να ξεκινήσουμε με τη σειρά από την κυρία Μαρινάκη. Thank you very much. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους ευρωβουλευτές για τις πολύ ουσιαστικές ερωτήσεις οι οποίες ενέπνευσαν όλους μας. Όσον αφορά τη μέθοδο εργασίας πρέπει να σας πω ότι προσπαθούμε να προχωρήσουμε συνεκτικά σε στενή διαδικασία με όλους τους συναδέλφους Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να υπάρχει αλληλοστήριξη μεταξύ μας και ε, είχαμε μία καλή κατανομή εργασίες μεταξύ μας, πράγμα το οποίο θα προχωρήσει για να μπορέσει να συνεχιστεί ο έλεγχος και η ισορροπία της εργασίας μας. Ε, υπάρχουν έγγραφα εργασίες και ενδεικτικά προγράμματα για την DCI, ε, MPF και ε, για την πυρηνική ασφάλεια και για τις ε, διαδικασίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε συνεργασία με την ΤΕΦΚΟ σχετικά με την ε, ανάπτυξη. Θα υπάρξει μία κοινή υποβολή απόφασης στο Κολέγιο των Επιτρόπων για υιοθέτηση και ε, θα υπάρξει και ε, χρηματοδοτητική βοήθεια την οποία θα παρακολουθεί η ΕΚΟ και η ΔΕΦΚΟ και θα πρέπει να προωθήσουμε και τις θεματικές ενότητες, ιδίως τις ε, ιδιαίτερες υπηρεσίες για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε τα θέματα για τον κύκλο του MMF σε συνεργασία με όλες τις υπηρεσίες ε, και του Κοινοβουλίου. Ε, όλα αυτά ενδιέφεραν ε, πάρα πολύ τα κράτη-μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ε, πρέπει γι' αυτό να συλλοθούμε στις ε, εξελίξεις της πολιτικής, στην οικονομική βοήθεια, ε, αποκλείοντας βέβαια την ανθρωπιστική βοήθεια, την στήριξη στην κοινωνία των πολιτών, που είναι τις εξωτερικές σχέσεις που είναι θέματα εκτός αυτού του πλαισίου. Και το Κοινοβούλιο εν ευθέτω χρόνο θα ικανοποιηθούν όσον αφορά την πρόσβαση στην αγορά, την οικονομική ανάπτυξη ε, και την ευξημένη κινητικότητα, ε, διευκόλυνση για τις θεωρήσεις και μεγαλύτερη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και όσοι ε, εταίροι δεν έχουν στηριχθεί θα πρέπει να ε, να ε, ε, εμπλακούν επίσης χωρίς όμως να τους τιμωρήσουμε. Θέλουμε να συνεχιστεί ένας διάλογος πολιτικός για να μπορέσουν να εποφεληθούν των εμπειριών που έχουμε αποκομίσει και θα χρησιμοποιήσουμε τα μέτρα αυτά για να αξιολογήσουμε την πρόοδο αλλά η αρχή more for more είναι νέα. Χρειάζεται μακροπρόθεσμη θεώρηση και δεν πρέπει να είναι μία απλή μηχανική άσκηση για όλους μας. Χρειάζεται ολιστική αντιμετώπιση και ε, θα πρέπει να συμβάλλουμε ε, όπως άλλωστε με τα χαρά θα περιμένουμε και τις δικές σας ε, επεμβάσεις. Για το θέμα της ε, ε, συνεργασίας των βορείων χωρών δεν θα επηρεαστούν, ε, θα υπάρξουν μέσα χρηματοδοτικά. Δεν μπορώ να σας πω ακριβώς στοιχεία τώρα, αλλά ίσως συνάδελφοι μπορούν να μας σας πούν κάτι παραπάνω, αλλά η βόρεια διάσταση παραμένει στο επίκεντρο των προσπαθειών μας. Όσον αφορά την EEAD, που ανέφερε η κυρία Μουνής δεν έχει ακόμη καταρτιστεί επισήμως σαν νομική οντότης αυτή και πρέπει να βρεθεί μία νέα μορφή διότι δεν θα ήθελα να προεξοφλήσω τι μορφή θα λάβει διότι υπάρχει ήδη ευρεία συμφωνία και θα πρέπει να ακολουθήσουμε την αρχή της προσθετικής συμμετοχής πράγμα το οποίο θα εξετάσουμε πολύ προσεκτικά για να εμπλέξουμε τους πάντες και όσον αφορά τις νέες προτεραιότητες με λιγότερα χρήματα είναι κάτι που απασχολεί όλους μας και ε, θα υπάρχει και στήριξη της Ευρωπαϊκής Ενώσεως με ε, ποσά που έχουν δεσμευτεί ε, για, αυτό το, για αυτά τα θέματα και που θα έχουν την αναγκαία στήριξη και παραμένουμε στη διάθεσή σας. Οι συνάδελφοι έχουν δυνατότητα να προσθέσουν λεπτομέρειες εάν το επιτιμούν. Ευχαριστώ. Ο κύριος παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να απαντήσω σε κάποιες από τις ερωτήσεις. Ε, νομίζω ότι κάποιες αφορούν όλα τα μέσα και κάποιες αφορούν πιο συγκεκριμένα το μέσο πρωταξιακής βοήθειας. Ε, κυρία Γκόμες, ε, υπάρχει ένα κοινό στοιχείο στα διάφορα μέσα, στους διάφορους μηχανισμούς και υπάρχουν ε, κάποιοι κοινοί εφαρμοστικοί κανόνες και διαδικασίες και τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το μέσο πρωτοεξιακής βοήθειας υπάρχουν συγκεκριμένοι τρόποι που αφορούν τη διαχείριση ή την βοήθεια που χαρακτηρίζουν μόνο το ΙΠΑ. Και αυτό θα αναφέρεται συγκεκριμένα στον εφαρμοστικό κανονισμό σε σχέση με το μέσο περιοδεξιακής βοήθειας. Πολύ σοβαρά άκουσα, όπως είπε ο κύριο Κράτσιν, σε ό,τι αφορά την προβολή της βοήθειάς μας και αυτό είναι ένας αγώνας ε, που δίνουμε εδώ και καιρό, γιατί είναι αλήθεια ότι οι άλλες χώρες καταρθένουν να έχουν πολύ μεγαλύτερη προβολή και μερικές φορές ε, με ένα επίπεδο βοήθειας το οποίο είναι χαμηλότερο από τις Ευρωπαϊκές Ένωσης. Επίσης, είναι αλήθεια ότι οι ιδιαιτερότητες ε, της βοήθειάς μας ε, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. Οικοδομούμε θεσμού σε μεγάλο βαθμό, παρέχουμε υποστήριξη στην ε, ανάπτυξη θεσμών, ε, σε ευθυγράμμιση με το κεκτημένο και αυτά είναι project τα οποία δυστυχώς έχουν ε, μικρότερη προβολή από μια γέφυρα ένα δρόμο και αυτό πρέπει να το λαμβάνουμε υπόψη. Αλλά θα προσπαθήσουμε στο ΙΠΑ 2 να εργαστούμε περισσότερο επί των κοινωνικών και οικονομικών εξελίξεων. Θα πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη προβολή εκεί και θα πρέπει και θα προσπαθήσουμε να προσδιορίσουμε συγκεκριμένες δράσεις για να αυξήσουμε την προβολή στον εφαρμοστικό κανονισμό. Υπήρξαν ε, κάποιες ερωτήσεις που σχετίζονται με το σύνδεσμο μεταξύ των βελτιώσεων της πρόοδου που έχει σημειωθεί ε, και των ε, των της κατανομής των κονδυλίων. Αυτό είναι ένα θέμα που θέλουμε να το ρυθμίσουμε με το νέο μέσο, με το νέο μηχανισμό και προσπαθούμε να αναπτύξουμε για κάποιες ιδέες σχετικά με την αποζημίωση για τις καλές επιδόσεις και για χώρες που τα πάνε πολύ καλά, παραδείγματο χάρη ως προς την πρόοδο ε, που σημειώνουν προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και ως προς τις μεταρρυθμίσεις, αλλά επίσης ε, και ανταμοιβή για συγκεκριμένου τομείς, για συγκεκριμένους κλάδους στο ιστορικό μιας χώρας και ελπίζουμε αυτό να μπορεί να προκαλέσει και κάποιο ανταγωνισμό μεταξύ των διάφορων Υπουργείων. η συνέπεια μεταξύ του κανονισμού IPA με τους λοιπούς κανονισμούς. Έχουμε συγκεκριμένα μέτρα στον οριζόντιο κανονισμό και θα συμπεριληφθούν και στους συγκεκριμένους εφαρμοστικούς κανόνες και θα προσπαθήσουμε να διασφαλίσουμε ότι αυτά τα οριζόντια στοιχεία καλύπτονται παρκώς παρακολούθηση της πρόδρου και αυτό αποτελεί τμήμα του κανονισμού στο άρθρο 2 του σχεδίου κανονισμού Αναφέρεται η πρόοδος προς την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων, η οποία αξιολογείται βάσει συγκεκριμένου αριθμού δικτών και ανέφερα μόνο μόλις το μακρύ κατάλογο που υπάρχει στον κανονισμό. Τώρα, ε, διαφορά μεταξύ καλής και κακής επίδοσης. Ε, θεωρώ ότι ε, ως συνέπεια αυτού που έλεγα πριν έρχεται, η αξιολόγηση που θα κάνουμε στην έκθεση πρόοδου θα είναι και ένα στοιχείο καθοδήγησης από τη δική μας σκοπιά. Προσπαθούμε να προωθήσουμε και το συντονισμό με τους υπόλοιπους δωρητές, ε, κυρίως σε ό,τι αφορά στο ότι ένα από τα στοιχεία του προγράμματος της βοηθειάς μας στα Δυτικά Βαλκάνια ε, συνεργαζόμαστε πολύ στενά με τα λοιπά πιστοτικά ιδρύματα, την Παγκόσμια Τράπεζα, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Νοικοδόμησης και Ανάπτυξης και άλλους διεθνείς οργανισμούς και τα εθνικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Έτσι λοιπόν διασφαλίζουμε ότι και θα έχουμε μία συνεκτική προσέγγιση σε αυτόν και σε άλλους τομείς. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Τώρα το λόγο έχει ο κύριος Ρούντιξ Σάουερ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Κόμες, Θέλω να επανέλθω σε αυτό που είπατε για την εναρμόνιση των μηχανισμών. Στη διαδικασία προετοιμασίας, και γι' αυτό και το κάναμε από κοινού, όλοι οι μηχανισμοί έχουν τώρα την ίδια δομή. Τις ίδιες αρχές, Τι ίδιε διατάξεις για τον προγραμματισμό και υπάρχει ένας εφαρμοστικό κανονισμό. Δηλαδή, κάναμε πάρα πολύ δρόμο προκειμένου να εναρμονίσουμε τους μηχανισμούς και με τον ενιαίο εφαρμοστικό κανονισμό θέλουμε ακριβώς να αποφύγουμε στις διαπραγματεύσεις οι προτάσει πάλι να αρχίσουν να αποκλίνουν μεταξύ του Όχι, εμεί θέλουμε να συγκλίνουν. Πετύχαμε δηλαδή σημαντική πρόοδο. Αυτό που λέτε τώρα για τη διαφοροποίηση είναι κάτι διαφορετικό από τη γλώσσα που χρησιμοποιούμε στον DCI. Εσείς λέτε διαφοροποίηση ανάλογα με τη συμπεριφορά των κυβερνήσεων. Το έχουμε ήδη κάνει. Ποτέ δεν στηρίζαμε οικονομικά χώρες με πολύ κακή διακυβέρνηση. Βέβαια μπορούμε να το συζητήσουμε ποιες είναι οι καλές και ποιες είναι οι κακές. Διαφοροποίηση πάντως υπάρχει και θα συνεχίσουμε να την κάνουμε τη διαφοροποίηση γιατί τι κριτήρια έχουμε, τις εκλογές, την ελευθερία τύπου, το κράτος δικαίου, την καταπολέμηση της διαφθοράς. Όχι, στην Αιθιοπία όχι. Σταματήσαμε την οικονομική στήριξη. Αντιδράσαμε δηλαδή στην κατάσταση εκεί. Για το αν θα συμπεριληφθεί στον προπολογισμό ή όχι. Ξέρετε ότι η Επιτροπή πάντα έλεγε ότι ήταν υπέρ το Αναπτυξιακό Ταμείο να, μπει, να είναι στον προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά είπαμε επίσης ότι μια που βρισκόμαστε σε περίοδο λιτότητας, το να βάλουμε τώρα το EDF στον προπολογισμό ελοχεύει κινδύνους. Δεν θέλω να πω περισσότερα γι' αυτό. Θα ήταν πολύ επικίνδυνο να προτείνουμε κάτι τέτοιο. Θα είχαν μειωθεί τα κονδύλια για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης, αν το είχαμε κάνει αυτό, φοβάμαι. Ο πρόεδρος τώρα ρώτησε κάποια πράγματα. Ιδιαίτερα για το EDF και παρά το γεγονός ότι δεν προτείναμε να μπει στον προπολογισμό, προτείναμε να γίνεται ο ίδιος βαθμός ελέγχου όπως και γίνεται και για τους άλλους μηχανισμούς και ας παραμένει εκτός προπολογισμού. Το κάνουμε δηλαδή επίσημα παρόλο που δεν υπάρχει επίσημα νομική βάση, αλλά προτείναμε να χρησιμοποιήσουμε ακριβώς ε, τα ίδια επίπεδα ελέγχου. Τώρα για το συνολικό ε, ποσό του δημοσιονομικού πλαισίου δεν θα σχολιάσω. Αλλά ξέρετε όμως ότι στο κεφάλαιο 4 έχουμε αύξηση. Υπάρχουν βέβαια ζητήματα που είναι σημαντικά εδώ για τις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης με άλλες χώρες, δηλαδή τι θα μπορούσε να τα απειλή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η αναπτυξιακή βοήθεια για μας ακριβώς είναι ένας τρόπος να καταπολεμήσουμε τις ρίζες του κακού. Και γι' αυτό και θέλουμε αναπτυξιακή βοήθεια σε αυτές ακριβώς τις περιπτώσεις, ώστε να αποφύγουμε τις τάσεις που μερικές φορές διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν σε ορισμένες χώρες. Αναφέρθηκε και το θέμα της μετανάστευσης. Και εκεί ισχύει το ίδιο. Τέλος, η αύξηση στο κεφάλαιο 4 που θεωρεί και ένας και μικρό, εξαρτάται πώς το βλέπει κανείς. Η συνολική αύξηση κατά 20% ενός κεφαλαίου είναι μια ιδιαίτερα θαραλέα πρόταση. Ορισμένοι θα λέγανε ότι ένα με 2% είναι ήδη θαραλέα πρόταση. Συζητήστε το με τους συναδέρφους σας στην Επιτροπή Προπολογισμών, αλλά 20% για αύξηση ολόκληρου τίτλου είναι κάτι πολύ σημαντικό. Τέλος για τον κύριο Σαλαφράγκα δεν προτείνουμε να μην χρηματοδοτήσουμε τη συνεργασία με τις χώρες της Λατινικής Αμερικής. Πρώτα απ' όλα, μιλάμε για εκείνες οι οποίες έχουν αναπτυχθεί αποτελεσματικά, έχουν θετική ανάπτυξη και εκεί προτείνουμε διαφορετική συνεργασία από ότι με εκείνες οι οποίες δεν έχουν καταφέρει την ίδια ανάπτυξη και για τις οποίες προτείνουμε να συνεχίσουμε την αναπτυξιακή συνεργασία. Συνολικά η Λατινική Αμερική θα πάρει το ίδιο ποσό αλλά με διαφορετικού είδους συνεργασία. Είναι κάτι διαφορετικό. Δηλαδή, εμείς δεν είπαμε να μειωθούν τα χρήματα που πάνε στις χώρες της Λατινικής Αμερικής, αλλά να αλλάξει ο τρόπος που συνεργαζόμαστε μαζί τους. Και αυτό γιατί κάποιες από τις χώρες αυτές έχουν εξελιχθεί πολύ. Αυτά. Θέλω να επανέλθω όμως και για το European Endowment. Εφόσον αυτό περιοριστεί στις γείτονε περιοχές, είναι μια καλή έδειξη για το πού έρχονται τα χρήματα. Αλλά όπως είπε και η κυρία Μαρινάκη, όσο δεν υπάρχει απόφαση, δεν μπορούμε να εντοπίσουμε την πηγή της χρηματοδότησης. Ο κύριος Μακ, επόμενος ομιλητής. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Για να επανέλθω στο θέμα το οποίο έθεσε η κυρία Μπράντερ, ίσως δεν είμαι πολύ σαφής. Αυτό που είδαμε είναι ότι το μπορούμε να βοηθήσουμε με το IFS ιδίως μετά από φυσικές καταστροφές π.χ. στην IT όπου μπορέσαμε να ρυθμίσουμε το θέμα της ασταθίας που δημιούργησε η φυσική καταστροφή αυτό συνάδει με ό,τι μπορεί να κάνει το πρόγραμμα ΕΚΟ και αυτό είναι το μήνυμα που θέλω να περάσω. Δεύτερον, σχετικά με την απάντηση στο ερώτημα που έθεσε η κυρία Μούνης Υπάρχουν ήδη διαφοροποιήσεις χρήσεως και εδώ σχετικά με το σωστό ποσοστό το οποίο πρέπει να αφιερωθεί ε, και πιστεύουμε ότι η πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα πρέπει ε, να καλύπτει το 65% των ε, επιγόντων περιπτώσεων και να μπορεί κατά αυτόν τον τρόπο να χρηματοδοτήσει επαρκώς τους δύο άλλους άλλους ε, στόχους, δηλαδή πρόβλεψη των διαμαχών και ε, επίλυση των κρίσεων και θέματα ασφαλείας, αλλά θα επανέλθουμε και σε αυτά τα θέματα. Και τέλος, για να απαντήσω στο ερώτημα του τι μπορεί να κάνει το PI, σε σχέση με τις ε, εξαγωγικές πιστώσεις που δεν είναι ο στόχος αυτού του ταμείου ε, είναι να διευκολύνει την πρόσβαση στην αγορά για ορισμένες εταιρείες ε, σε συνεργασία με τις ε, εμπλεκόμενες χώρες για την κατάργηση των εμπορικών φραγμών και για την αύξηση της κινητικότητας. Αυτά είναι τα στοιχεία που περιέρχονται σε αυτό το θέμα. Σας ευχαριστούμε για αυτές τις ε, πλήρεις ε, τεχνικές και εξαντλητικές ε, παρεμβάσεις. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω να υπενθυμίσω ότι η προθεσμία για τις τροπολογίες είναι η 5η Ιουνίου στις 12 το μεσημέρι. Πιστεύω ότι δεν ζητά κάποιος άλλος το λόγο. Και πάλι σας ευχαριστώ όλους σας. Grazie, arrivederci. Είστε Colleghi, l'ultimo passo. Αγαπητοί λοιπόν, να περάσουμε στο τελευταίο στάδιο. Λίγη ησυχία σα παρακαλώ, γιατί πρέπει να συνεχίσουμε τις εργασίες μα. Έχουμε το τελευταίο σημείο, ηλεκτρονική ψηφοφορία για τον ορισμό μια νέα συνεργασία με τη Λατινική Αμερική. Η κυρία Αντρική Ένε είναι η η συγγήτρια, της γνωμοδότησης. Έχετε την κάρτα για να περάσουμε στην ψηφοφορία. Είναι. Ωραία. Τροπολογία 1. Με προφορική τροπολογία υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 2 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Προφορική τροπολογία υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 3 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία προφορική 3 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Προφορική τροπολογία 4 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 4 υπέρ. Αποχές. Κατά διορθώνει ο πρόεδρος. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία. 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 7. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 8. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 9 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 10 Έχουμε τμηματική ψηφοφορία, πρώτο τμήμα, ποιος είναι υπέρ. Κατά, αποχές, απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα, υπέρ. Κατά, αποχές, απορρίπτεται. Προφορική τροπολογία 5, υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 11. Όχι. Καταπίπτει. 12. Επίσης. 13. Τροπολογία 13 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Προφορική τροπολογία 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 14. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Υπορρίπτεται. Τροπολογία 7, προφορική υπέρ, κατά, εποχέ, εγκρίνεται. 8, προφορική τροπολογία υπέρ, κατά, εποχέ, εγκρίνεται. Τροπολογία 15, υπέρ, κατά, εποχέ, εγκρίνεται. 16. Λοιπόν, περνάμε στη 17. Προηγούμενη καταπίπτη, υπέρ, κατά, εποχές, εγκρίνεται. 18 υπέρ. Κατά. Οχές. Απορρίπτεται. Για τα 19 υπάρχει έτοιμα προφορικής ε, τροπολογίας από την κυρία Αντρικίνε. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Έχω μια προφορική τροπολογία. Το κείμενο λοιπόν ε, θα έλεγε ότι, ότι την ε, είπατε εκπρόσωπο, αντιπρόεδρο της Επιτροπής, ε, να διαβουλευτεί και να ενημερώσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το εφιστάμενο διάλογο για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα λοιπά, όπως το βλέπετε στο κείμενο. Σας ευχαριστώ. Υπάρχει αντίρρηση. Παρακαλώ κύριε Σαλφράγκα. Καμία αντίρρηση, να ψηφίσουμε. Υπέρ κατά, εποχές, εγκρίνεται. Λοιπόν, να περάσουμε στην ψηφοφορία του κειμένου στο σύνολό του υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονική ψηφοφορία. Μάλιστα, λέει ο πρόεδρος. Ηλεκτρονική ψηφοφορία. Άρχεται η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ancora κολέγα Ένας ακόμη συνάδελφος. Πέρας. Λοιπόν, εγκρίνεται με ευρία πλειοψηφία. Σας ευχαριστώ για τη συνεργασία. Υπάρχει η ψηφορία.